pääohjelmaan ja sanon vain lyhyesti, että meillä on Εγώ. Eh, Θέλω να κάνω μερικές ε, ανακοινώσεις προτού προχωρήσουμε στο πρόγραμμα ε, διότι έχουμε εδώ τον κύριο Άλεξ Βαν Νόβελ, ε, τον οποίον καλωσορίζω, διότι θα μιλήσει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι κάτι που παρακολουθούμε πολύ εκ του και μετά θα συζητήσουμε την έκθεση του κοινίου Κούκα που, που πραγματεύεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Καταρχήν όμως θέλω να σας πω ότι είναι 20 χρόνια από όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Όλοι πρέπει να ξεχνάμε αυτή την... αυτό το γεγονός και τη σημασία του για τα ανθρώπινα δικαιώματα διότι ήταν ε, η πτώση της Δυτικής Γερμανίας ε, ο λαό αυτός απέκτησε δικαιώματα υπάρχει ακόμη ένας αόρατο στίχος που χωρίζει την Ανατολική από τη Δυτική Γερμανία αλλά έχει καταρρεύσει η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας ε, και αυτό συνέβη χωρίς να χυθεί μία σταγόνα αίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε δύο μέρες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε μία εκδήλωση επίσημη όπου θα συζητήσουμε τα γεγονότα στην ε, ε, Ανατολική Γερμανία πριν 20 χρόνια θα καλέσουμε και νέους που γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 1989 από διάφορα κράτη για να συζητήσουν με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τον κύριο Μπούζεκ και τους αντιπροέδρους για το ρόλο και τη σημασία του Κοινοβουλίου για αυτούς. Η συνεδρίαση λοιπόν αυτή είναι στις 10 ε, ε, και στη συνέχεια ε, στην αίθουσα Α3G3 και συνέχεια ο κύριος Μπούζεκ θα μία εορτή για τα γεγονότα που, θα, που έλαβαν χώρα πριν 20 χρόνια και θα αναφερθεί στην ελεύθερη Ευρώπη του 1989. Θα παρουσιαστεί και ο, ο Τσέχος πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βάσλαφ Χάβελ και στη συνέχεια θα έχουμε μία επίσημη ε, τελετή πριν ξεκινήσει η μίνι ολομέλεια. Θα μιλήσει και ο Βάσλαβ Χάβελ και ο πρόεδρος κύριος Μπούζεκ. Αυτά είχα να σας πω για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα. Θα ήθελα να σας πω επίσης ε, ε, σχετικά με άλλα γεγονότα που είχαν λάβει η χώρα από τις τελευταίες συνεδρίασεις μας ότι έχουμε την δυνατότητα να, να συζητήσουμε με την Αμερικανική Διοίκηση, με τους εκπροσώπους της Αμερικανικής Πρεσβείας και φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να δεχτούμε εδώ τον νέο εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κύριος Μπόσνερ ε, είναι ε, ο οποίος έρχεται από την μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights First. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ένας από τους στόχους μας είναι να στείλουμε του χρόνου μία μικρή αντιπροσωπεία στη Washington. Ίσως θυμάστε ότι ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του τους οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ήρθε να μας ε, επισκεφθεί στο Στρασβούργο. Ο κύριος Αγγίλα, ο πρόεδρος και εγώ ε, κληθήκαμε για μία ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτά θα διεξαχθούν στο Στρασβούργο στις 23 Νοεμβρίου και ε, θα συζητήσουμε με τους διάφορους εκπροσώπους από το Συμβούλιο της Ευρώπης όπου τα πράγματα είναι πολύ εξελιγμένα και γίνονται σοβαρές συζητήσεις και ενδέχεται ο πρόεδρος να επανέλθει να ξανασυζητήσουμε στους επόμενους μήνες. Ε, πήγα επίσης στη Χάγη και βρήκα όταν ε, πάρα πολύ σημαντικό να συναντήσω τον πρόεδρο Σόγκ και την ε, κυρία Φάτο Μπενσούντ, την ε, την αναπληρώτρια εισαγγελέα και τους ανέφερα ότι στηρίζουμε τις εργασίες του ποινικού δικαστηρίου όχι μόνο ηθικά αλλά και ουσιαστικά. και του χρόνου θα γίνει στην Ουγκάντα μία διάσκεψη και θα καλέσουμε πριν από αυτό τον πρόεδρο Σόγκ για να μπορέσει να ε, συζητήσει μαζί μας περί τίνος πρόκειται να πραγματευτεί ε, αυτή η ε, διάσκεψη ήρθαν και ε, Ρώσοι εκπρόσωποι εδώ οι οποίοι μας ε, επέδωσαν ένα τεράστιο έγγραφο σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και είχαμε σκεφτεί ότι όντως έπρεπε να γίνει ε, κάτι σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία. Αυτό βέβαια είχε συζητηθεί μόνο άτυπα με ε, τον αντιπρόεδρο του δικαστηρίου. Συζητήσαμε επίσης ε, για την ε, συζήτηση του κυρίου Μπασία στην Τουρκία όπου αναφερθήκαμε στην στήριξη ε, των της Ευρωπαϊκής Ενότητας στην ICC και όλα αυτά είναι γεγονότα για να δείξουμε τη στήριξη την οποία παρέχουμε στην ICC. Κατά τρόπον να μπορέσει να προσαχθεί ο κύριος Μπασίρ στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο. Ο κύριος Κάζακ ήθελε κάτι να προσθέσει σχετικά με την διακυβερνητική συζήτηση με την Τουρκία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ήθελα να σας παρουσιάσω τα προσωπικά μου συμπεράσματα και στη συνέχεια στη συνέχεια της συναντήσεως η οποία έγινε στην Άγκυρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας και ε, συγκεκριμένα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις διότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Τουρκία και τις χώρες των, των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ε, δημοσιευθεί. Το ίδιο ισχύει και ε, για την ε, συζήτηση της διεύρυνσης κατά το 2009-2010. Συζητήσαμε όντως όλα αυτά τα θέματα με τους Τούρκους συναδέλφους μας και ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών κριτηρίων προσβλέποντας προς μία προσχώρηση και την ε, ε, ε, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε με τα ικανοποιήσεως της εξελίξης και την πολιτική του Πρωθυπουργού προς, προς ένα δημοκρατικό άνοιγμα, μεγαλύτερη διαφάνεια ε, μία πιο ευρεία συζήτηση των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν ε, από πολλού αλλά που δεν έχουν συζητηθεί δημοσίως. Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει εις ε, τους, τους αντι καθεστωτικούς Κούρδους να μπορέσουν να επιστρέψουν δηλαδή ε, υπάρχουν ε, διάφορες, ε, διάφορα κινήματα κουρδικά ένα εμφύλιος πόλεμος ο οποίος απλώς έχει πολλά θύματα και γι' αυτό σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι έχει ξεκινήσει ένας διάλογος με τις διάφορες διάφορες ε, θρησκευτικές μειονότητες ιδίως όσον αφορά τις ιδιοκτησίες των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων και συγκεκριμένα των χριστιανικών. Έχουμε εκφράσει τη στήριξή μας κατόπιν των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί προς ε, ε, μία ε, ομάδα μέσων ενημέρωσης τουρκικής διότι υπάρχει περιορισμός ε, τη ελευθερίας του τύπου και του λόγου και οι συνάδελφοι ε, επίσης έθιξαν το θέμα της ισότητος ε, αντιμετωπίσεως των ανδρών και των γυναικών και επεσήμαναν ε, τα δικαιώματα ορισμένων ευάλωτων ομάδων όπως οι ε, ομοφιλόφιλοι και άλλοι αναφερθήκαμε στα συνδικαλιστικά δικαιώματα ή στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε όλα τα προβλήματα αυτά ε, αναφέρθηκαν επιμείναμε και προσπαθήσαμε να να αναφερθούμε ε, σε στα δικαιώματα του ανθρώπου χωρίς όμως να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ε, υπήρχε, υπήρχαν ορισμένες διαφορές ε, με τους Τούρκους ομολόγους μας ε, και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε μια κοινή ανακοίνωση κύριε Πρόεδρε και αυτά ήταν τα προβλήματα όπως προέκυψαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάτζακ για την... Ε, αν ήταν εδώ ο κύριος Σόμπιλ θα μπορούσε επίσης να σχολιάσει σχετικά με την ε, έκθεση ε, των εξωτερικών υποθέσεων στη Μαδρίτη, αλλά τυχώς δεν έχει έρθει ακόμη. Μήπως μπορώ να σας παρακαλέσω να έχετε λίγη υπομονή, διότι συνέβησαν τόσα πράγματα την Παρασκευή Όλοι στο Κοινοβούλιο είχαμε μια πολύ σημαντική ημέρα, μάλλον θα έχουμε ε, μια σημαντική ημέρα, διότι ε, θα έχουμε ε, την ακρόαση του του μελλοντικού επιτρόπου είναι πολύ ε, σοβαρό θέμα και αυτό θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου η ακρόαση αυτή δηλαδή. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το Ουσμπεκιστάν και ε, τέλος Οκτωβρίου η οι Υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν να άρουν ε, το εμπάργο οπλισμών ε, προς το Ουσμεκιστάν, συζήτησαν με ε, τις αρχές και συμφώνησαν ότι πρέπει να δώσουν και επιπλέον σήματα ενδείξεις καλής θελήσεως διότι πρέπει να σκεφτούμε τι μέτρα ακόμη θα χρειαστούν προς το Ουσβεκιστάν διότι αφενός έρεται το εμπάργο πλεισμών αλλά έχουμε πολλά προβλήματα με το Ουσμπεκιστάν και θα πρέπει να καλέσουμε το Ουσμπεκιστάν να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Σχετικά με το επόμενο θέμα, είχαμε μία ενδιαφέρουσα επίσκεψη από τη Βόρειο Κορέα. Και αυτό ήταν ε, ε, ε, σχετικά με τα θύματα των στρατοπέδων της Christian Solidarity και ακούσαμε πολλούς μάρτυρες σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς που υπάρχει εκεί. Ε, του χρόνου θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την περίπτωση της Βορείας Κορέας και να καλέξουμε τον Βέτεκ ε, Βούντερ Μπράουν εκπρόσωπον του ΟΗΕ ε, για την περιοχή εκεί να έρθει να συζητήσουμε να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την ICC και πώς μπορούν να λειτουργήσουν εκεί οι διεθνείς οργανώσεις. Το επόμενο θέμα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα στη Στοκχόλμη υπήρξε ε, μία συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ρωσίας και θα ενημερωθούμε περί των τελευταίων εξελίξεων που μπορεί ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ότι η αντιπολίτευση ε, έχει ε, πάλι ένα θύμα τον κύριο Μάσρεπ ο οποίος ε, δολοφονήκεται και 4 Οκτωβρίου άρα θα πρέπει όντως να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους κυρίους αυτούς διότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσμενής την εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε πολλά. Θα δούμε τον κύριο Μιλίκεβιτς, ο οποίος είχε, ε, είχε πάρει το βραβείο Ζαχάροφ του 2006. Ε, θα έρθει εδώ στη συνεδρίασή μας ε, του Νοεμβρίου 30 Νοεμβρίου δηλαδή και ε, ήθελε να συναντηθεί οπωσδήποτε με τους εκπροσώπους της Επιτροπής μας. Δεν ξέρω εάν έχω να σας πω κι άλλα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορα ψηφίσματα από το Κοινοβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση. Ε, μπορώ ίσως να αναφερθώ στην κατάσταση στη Γουινέα και σχετικά με την επίσημη γραμμή αναμένουμε ότι αυτή η ε, πολεμοχαρής χούντα θα συνεχίσει να διοικεί την ε, Γουινέα και ε, γι' αυτό είχαμε προσφάτως τόσα πολλά θύματα. Ξέρουμε ότι ακόμη και τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται εκεί και χρειάστηκε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να δραπετεύσει διότι δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει εκεί. Ε, αυτά είχα να σας πω. Μπορώ έτσι να κλείνω, κλείσω αυτό το θέμα και να φτάσουμε τώρα στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου ε, εξετάζουμε τις εξελίξεις ε, στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στον ΟΗΕ και θέλω να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Άλεξ Βαν Μεβεν ο οποίος σαν εκπρόσωπος του Βελγίου ηγείται αυτής της αντιπροσωπείας ε, θέλω να καλωσορίσω και τους άλλους παρισταμένους από την ίδια οργάνωση. Έχουμε εδώ τον ε, τμήματάρχη ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Θέλαμε τη συζήτηση αυτή να την κάνουμε ήδη τον Οκτώβριο, αλλά ο κύριος Βαν Μέμπερ δυστυχώς είχε εκείνη την εποχή να διεκπαιρεώσει πιο σοβαρά θέματα και υποθέτω ότι αυτό θα συζητηθεί και εδώ. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε καλές και ενεργές σχέσεις με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γι' αυτό και στέλνουμε ε, συχνά μία αντιπροσωπεία εις ε, το Συμβούλιο αυτό. Ήθελα να σας πω ότι τον Ιανουάριο είχαμε υιοθετήσει την έκθεση Αντρικένε σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ρόλου των ανθρω... της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά τα στοιχεία τα έχετε στο υλικό που σας έχουμε στείλει και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Βαν Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται να μπούμε σε άμεσο διάλογο με τα μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως Προέδρου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να μοιραστώ μαζί σας την άποψή μου για τις δραστηριότητε του Συμβουλίου αυτού. Αναγνωρίζουμε την ε, συνεχιζόμενη, ε, το, το μόνιμό σας ενδιαφέρον και δραστηριότητες για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία αυτών, καθώς και για την προστασία των βασικών ανθρώπινων ελευθεριών. Ε, προεδρεύοντας ε, του βασικού ως όργανου των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τιμή μου αλλά και καθήκον να εργάζομαι όχι μόνο για τη νέα το νέο διακυβερνητικό σώμα αλλά και για να πληρωθούν οι προσδοκίες πολλών παρατηρητών από τη δημιουργία του, από, τη γενική, από το ψήφισμα μάλλον 60 κάθετος 251 ε, στις 15 Μαρτίου 2006 με το ψήφισμα δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει προχωρήσει πολύ, έχει φτάσει σε ένα δεσμευτικό πακέτο που καθοδηγεί τις εργασίες του και οδήγησε στον εξορθολογισμό και την ε, καλύτερη διαχείριση. Έχουμε τακτικές ε, συνόδους, συζητούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε μπει σε διάλογο με διάφορους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονε ε, καθώς και έχουμε φτιάξει διάφορα, έχουμε μάλλον ε, αντιμετωπίσει διάφορες κλιμακούμενες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον πολλέ χώρε έχουν εθελοντικά περάσει από την νέο καθολικό μηχανισμό εξέτασης ε, συμπεριλαμβανομένων 11 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο χρειάστηκε να αποδείξει την ικανότητά του να, να... να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μόλις έρχομαι από τη Νέα Υόρκη όπου παρουσίασα μια έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την Γενική Συνέλευση και μπορούμε να πούμε ότι κατά το έτος 2008-2009 οι προσπάθειές μας ήταν καρποφόρες ε, όσον αφορά την επιχειρησιακή μας απόδοση αλλά και ως προς τις ε, δυνατότητες για καινοτομία και εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα θα ε, ήθελα να σας δώσω μια πιο ε, συγκεκριμένη άποψη για τα επιτεύγματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ολοκλήρωσε τι εργασίε του τον Οκτώβριο του 2009. Ήταν η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να προεδρεύσω τον, τη τακτική του Συμβουλίου και ήταν πραγματικά τρει ε, πολύ ε, έντονες εβδομάδες, αλλά νομίζω πως τα αποτελέσματα ήταν γενικά θετικά. Κατά τη διάρκεια των 12 συνόδων το Συμβούλιο συζήτησε για διάφορες ε, εκθέσει υψηλού επίπεδου και ξεκίνησε διάλογο με ειδικέ διαδικασίες ε, όπως για παράδειγμα τον ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά σε ένοπλες σειράξεις ή τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σομαλία. Το Συμβούλιο έκανε επίσης συζητήσεις σε πάνελ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών στα κέντρα κράτηση καθώς και για την σωμάτωση της προπτικής ε, των διαφορετικών φύλων ε, στις διαδικασίες μετανάστευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην, ε, στις συγκριτικές εκθέσεις που γίνονται για τις διάφορες χώρες. Θα ήθελα να τονίσω τους εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν για να εξετάσουν την, ανθρώπινη, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν και τα πολιτιστικά δικαιώματα αντίστοιχα, καθώς και την παράταση της εντολής για την Σομαλία και την στην Καμπότζη και τη συνέχιση της εντολής για τον Μπουρούντι. Το Συμβούλιο επίσης έλαβε μια ενημέρωση από τον ΥΠΑ, Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Μαρή Πιλάρ, για θέματα δικαιωμάτων που εξακολουθούν να ανησυχούν την κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ένα ψήφισμα για την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Βυρμανία, Μιανμάρ, που υιοθετήθηκε ομόφωνα και υποστήριξε την πρωτοβουλία της των χωρών της Λατινικής Αμερικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ονδούρα. Τα μέλη και οι παρατηρητές συζήτησαν μια έκθεση της, ε, αντιπροσωπείας, της αποστολής μάλλον ανέβρεσης στοιχείων, της οποίας ηγήθηκε ο Ρίτσαρντ, Ρόσαν, ξεκινώντας ε, διαδραστικό διάλογο με όλα τα μέλη αυτής της αποστολής και υιοθέτησε ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα πελαστανιακά εδάφη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 ειδικών συνόδων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα, το θα συνεχίσει να παρακολουθεί την έκθεση ντόσων ε, κατά τις 13η Σύνοδό τον επόμενο Μάρτιο. Ω τμήμα τη περιοδική καθολική έκθεση, 16 ακόμα εκθέσει υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια τη Συνόδου του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων εκείνε που αφορούν το Αφγανιστάν, το Βανουάτου, τη Χιλή, το Βιετνάμ και την Ιεμένη. Το κλείσιμο της Συνόδου ε, βρήκε συγκεκριμένα 41 κείμενα που αφορούσαν διάφορα θέματα. Να σας αναφέρω ψηφίσματα για την ελευθερία έκφρασης, τις διακρίσεις κατά των γυναικών και ένα που αφορά το πόσιμο νερό και την υγειονομική κατάσταση. Για να σας αναφέρω μόνο λίγα από αυτά. τα μέλη του Συμβουλίου υιοθέτησαν ε, ε, συνενετικά ένα ψήφισμα που, καθισ... που ένα μια διακυβερνητική ομάδα που στόχο θα έχει τη βελτίωση της λειτουργίας του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ζήτησε να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις σχετικά με τη διαδικασία της αναθεώρησης πριν από την ε, συνέλευση της ομάδας αυτής που θα γίνει στο πρώτο ήμεση του 2010 θα εστιάσουμε τις ε, συζητήσεις μας σε σχέση με τη δικασία αναθεώρησης για θέματα, σε θέματα διαδικαστικά. Εγώ στόχο έχω να υποβάλω προτάσεις ε, σύμφωνα με το ψήφισμα 251 κατά το δεύτερο ήμιση της ε, εντολή μου και στόχο θα έχουν να διευκολύνουν τις συζητήσεις για το θέμα αυτά, αυτό και την επίτευξη συνένεσης για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε Πράγμα που θα γίνει με το διάδοχό μου τον επόμενο χρόνο. Σκοπεύουμε να λάβουμε υπόψη τις απόψεις ε, των, ε, όλων των ενδιαφορεμένων φορέων. Ενώ συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την ατζέντα μας και τις μεθόδους εργασίας μας, η διαδικασία εξέτασης των διαφόρων εργασιών δεν θα σταματήσει, ούτε και η εφαρμογή των, ε, της κοινώς συμπεφωνημένης εντολής. αυτό θα, αυτό θα το μερινήσω ιδιαίτερα να γίνει και θα ε, καλέσω όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, στόχο έχει να εκτελέσει την εντολή του όπως ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά ε, υπό διαφορετικές μορφές και ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων ε, που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζω πως παρακολουθείτε στενά τις εργασίες του Συμβουλίου και ότι έχετε εξαίρετη γνώση των μηχανισμών του και των επιτευμάτων του μέχρι στιγμής. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την έκθεσή σας για την εξέλιξη του Συμβουλίου καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Τη 3ης Ιανουαρίου 2009. Επίσης γνωρίζω πως ε, ορισμένες φορές απογοητευθήκατε από την απόδοση του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που με προσφέρετε σήμερα για να ανατρέξουμε κάπως στο τι έχει γίνει και να εξετάσουμε το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο για να βρούμε δικαιολογία στα θέματα που θα μπορούσε να έχει ενεργήσει πιο αποτελεσματικά, αλλά για να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ε, μπορέσαμε μπορέσαμε πάντοτε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Ε, καλύτερη κατανόηση θα μας επιτρέψει, πιστεύω, να ε, επωφεληθούμε τα μέγιστα των ε, δυνατοτήτων που υπάρχουν για βελτίωση της απόδοσης του Συμβουλίου στην άσκηση της εντολής του και να ανταποκριθούμε περισσότερο στις προσδοκίες που έχουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα θύματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον Μάιο του 2006 να δημιουργήσει το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να του αναθέσει το έργο να προωθήσει άνευ καμίας διάκρισης την καθολικό σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα κράτη-μέλη τότε είχαν ε, δικρουόμενες απόψεις όσον αφορά το, τη θέση που θα έπρεπε να κατέχει το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ε, δομών του ΟΗΕ και για τα μέσα τα οποία θα έπρεπε να έχει στη διαθεσή του για να μπορέσει να εκτελέσει την εντολή του. Αυτές οι αντικρουόμενες απόψεις των κρατών μελών που πολύ συχνά ε, συγκεντρώνονταν σε περιφερειακή βαθμό επηρεάζουν ακόμα τη ε, λειτουργία του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν καταφέρνουν πάντοτε να συμφωνήσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πληρεί το ρόλο του το Συμβούλιο απέναντι στην θέσπιση προδιαγραφών, την εποπτεία ή την τεχνική αρρωγή σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορώ παρά να σα επιβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν λειτουργεί εν κενό. Οι καθημερινέ πραγματικότητε, οι κοινωνικέ, πολιτιστικέ, οικονομικέ και πολιτικέ διαφορέ ανάμεσα στα κράτη και τι ομάδε κρατών επηρεάζουν τι εργασίε αυτού του διακυβερνητικού οργάνου. Τα θέματα, τα ερωτήματα μάλλον που θα πρέπει να θέσουμε είναι τα εξή. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη να μην ξεχνούν την εντολή του Συμβουλίου. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το Συμβούλιο θα χρησιμεύσει ως ένα φόρουμ για διάλογο για θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν επικοδομητικά όλους τους μηχανισμούς του Συμβουλίου. Πώς μπορούμε να πείσουμε τα κράτη πως η εποπτεία η παρακολούθηση και ο εντοπισμό ε, συγκεκριμένων προκλήσεων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συμβαδίζουν με τον ορισμό και την παροχή μια αρρωγή, είτε αυτή είναι τεχνική φύση είτε άλλη φύση. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να βρούμε την αρχή στις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα το, εκτός από το, για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπεύθυνο και για τα διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα. Δεδομένου στις περιορισμένες εντολής είμαι προσιλωμένος στην, στην ανάληψη των ευθυνών μου και στην διεξαγωγή επικοδομητικού διαλόγου για όλα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θα υποστηρίξω κάθε προσπάθεια που ε, θέλει να τοποθετήσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ατζέντα του Συμβουλίου ε, χωρίς ε, να έχω επιλεκτικές ε, διαθέσεις. Είμαστε ένα καθολικό όργανο, όπως καθολικά είναι και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως έχω, δηλώσει σε πολλές ευκαιρίες, ε, είμαι δεσμευμένος στο να να, να βοηθήσω στην οικοδόμηση ε, γεφυρών, γεφυρωμάτων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες. Επίσης, θέλω να μεριμνήσω για την ανακαιρεότητα και την ανεξαρτησία των ειδικών διαδικασιών. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει διάφορους μηχανισμούς στη διάθεσή του, και ο καθένας έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία. Εγώ θεωρώ πως είναι καθήκον μου να βοηθήσω να διασφαλιστεί η πλήρης χρήση και σεβασμός των διαφόρων ε, διαδικασιών λειτουργίας κάθε μηχανισμού προς όφελος της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του Συμβουλίου. Επιπλέον, έχω δεσμευθεί στο να διασφαλίσω την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της εργασία του Συμβουλίου. Από τον διορισμό μου έχω έρθει σε επαφή με εκπροσώπους των ΜΚΟ και των εθνικών ε, θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τακτικό ρυθμό. Αξιολογώ, αξιοποιώ τις απόψεις τους και είμαι πεπισμένο για τον απαραίτητο ρόλο τους στο να θυμίζουν στα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους στα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διασφάλιση και την πλαισίωση των εργασιών του Συμβουλίου. Είναι κάποια αυτά παραδείγματα της προσπάθειας για την αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και επικοδομητική δέσμευση με τους μηχανισμού του. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είμαι πεπισμένο ότι είναι απαραίτητο ο ρόλο του νέου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντό ε, τη ευρύτερη κοινότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό με στόχο την καλύτερη προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, θεμελιωδών ελευθεριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, λαμβάνοντα υπόψη όχι μόνο αυτή την εντολή, αλλά Επίσης, τα βασικά της χαρακτηριστικά, καθώς και τον κόσμο εντός του οποίου λειτουργεί, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις ελπίδες ταυτόχρονα. Η δουλειά μας στη Γενέβη μπορεί μόνο να ωφεληθεί από ρεαλιστικές προσδοκίες πρέπει να συνεχίσουμε και να διασφαλίζουμε όχι μόνο τη σωστή χρήση και την ενίσχυση των μηχανισμών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά επίσης ε, την ε, σωστή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα του ΟΗΕ καθώς και οι οργανισμούς αυτού. Σας καλώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσετε να στηρίζετε την εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών υπό τη διεθνή νομοθεσία, το διεθνές δίκαιο. Επίσης θα ήθελα να σας καλέσω τακτικά να θυμίζετε στους συναδέλφους ε, σε τρίτες χώρες ε, για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει αυτές οι ίδιες όταν έγιναν μέλη του Συμβουλίου τις συστάσεις που γίνονται προς τις χώρες αυτές μέσω της διαδικασίας UPR καθώς και την ανάγκη να συνεργαστούν με τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου θεωρούμε ότι είναι δέσμευσή μας να είμαστε πολυμερείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει πρόσβαση στις άλλες, ε, ε, ε, όχι μόνο στα κατημέλη, αλλά και σε άλλες περιφερειακές πολιτικές ομάδες, ώστε να εξηγεί τις θέσεις της, αλλά και τις ανησυχίες της. Χρειαζόμαστε επίσης την υποστήριξή σας, ώστε να έχουμε το στένος να προβούμε σε επικοδομητικό διάλογο για τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ για την, για την προσοχή σας. Eh, Ευχαριστώ πολύ τον πρέσβη κύριο Φαν Μεύεν. Προσπαθήσατε να ακολουθήσετε και κάποιες βασικές συστάσεις ε, των δικών μας ψηφισμάτων και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να προσβλέπουμε στην, στο μέλλον σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον τμήματάρχη από το γραφείο του είπα του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Υποεπιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μπορώ να λάβω μέρος σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη συζήτηση αυτή Δεν να χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και με μεγάλη ε, χαρά ε, προσβλέπω στη συνεργασία με την υποεπιτροπή σας. <clears throat> Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω ε, τον, την παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, με τον οποίο σίγουρα θα συνεργαστούμε. Όσον αφορά την ε, στήριξή μας στη λειτουργία του Συμβουλίου, το να κινηθεί κανείς από την, από από την Κομισιόν, στο Συμβου... από την Επιτροπή μάλλον στο Συμβούλιο, δεν ήταν πολύ εύκολη περίπτωση. Υπήρξαν πολλές εντάσεις, ε, γιατί δεν ήταν όλοι διεθνώς υπέρ της πολυμερούς σε Διάφορες ε, πρωτοβουλίες ξεκίνησαν ώστε το 6251 να είναι επιτυχές, το ψήφισμα που ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος, να είναι επιτυχές, να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις χωρίς όμως να υπονομευθούν τα όσα ήδη υπήρχαν. Με αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα, ο ρόλος του Συμβουλίου και η προστασία, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζεται σε διεθνή φόρα ε, με νέα σύνθεση είμαστε ψηλότερο ε, στάτους και καλύτερη ευχέρεια, μεγαλύτερη ευχέρεια για τη σύγκληση ειδικών συνόδων. Η καθολική σύγκριση αποτελεσμάτων είναι ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα, μεγάλα επιτεύγματα του Συμβουλίου μέχρι στιγμή, Με αυτό το νέο μηχανισμό όλα τα κρατημέλη υποβάλλουν μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτή μετά συζητείται από το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση και συνδέεται με δύο εγγράφα τα οποία προετοιμάζονται από την ε, υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από ΜΚΟ και από τα ειδικά όργανα του ΟΗΕ, ειδικού ε, εισηγητέ και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμή το Συμβούλιο έχει εξετάσει 80 τέτοιες εκθέσεις και το UPR ε, είναι μια διαδικασία που έχει προχωρήσει ως ένα βασικό επίτευγμα του Συμβούλου αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα όσον αφορά την υποβολή τέτοιων ε, γραπτών εκθέσεων. Ε, έχουμε αντιπροσωπήσει ακόμα και από μικρές χώρες όπως το Βανουάτου που άνθρωποι που έρχονται από ολόκληρο τον κόσμο για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, στις αποστολές μάλλον στη Γενέβη. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή των Τρόικα, αυτών αποτελούμε εμεί Τρόικα, μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών και των κρατών παρατηρητών ε, όσον αφορά τα κράτη που είναι υπό εξέταση. Το Συμβούλιο επίση έχει δείξει σημαντικά δείγματα ευελιξία όσον αφορά την εξέταση των θεμάτων, ε, συγκαλώντα ειδικέ ε, συνόδους. Έχουμε μέχρι στιγμής 12 τέτοιε ειδικέ συνόδου και προσαρμόζοντα την οργάνωση πάνελ ο χώρος που δίδεται στις ειδικές διαδικασίες, αυτό που αποτελούμε κοσμήματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει αυξηθεί και περισσότερος χρόνος και χώρος παρέχεται σε αυτές. Η διάδραση με τον Υπατοαρμοστή ε, που αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Πρόεδρο έχει επίσης επεκταθεί, είναι καλύτερα δομημένη, γίνονται τακτικές ε, ενημερώσεις, ε, σχόλια και συμμετοχές των αποστολών και πολυάριθμες ευκαιρίες για τον είπα να παρουσιάσει τις εκθέσεις και τα σχόλιά του. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου του Σεπτεμβρίου, ο ύπατος αρμοστής ενημέρωσε το Συμβούλιο για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 42 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όσον αφορά την Ευρώπη, η σημαντική είναι η κατάσταση των Ρώμα σε διάφορες χώρες, καθώς και η αντιμετώπιση των μεταναστών. Αυτό σημαίνει πως το Συμβούλιο λειτουργεί στο μάξιμουμ των ικανοτήτων του και δεν υπάρχει χώρος για βελτίωση. Φυσικά και όχι. Όπως οποιαδήποτε άλλη δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο αντιμετωπίζει προκλήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ε, περιοδικής ε, επανεξέτασης που θα γίνει σύντομα. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε θέματα όσον αφορά το καθεστώς του Συμβουλίου που είναι καταρχήν ευθύνη των μελών του που αποφασίζεται στο επίπεδο της ε, γενική συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Όποια και αν είναι τα συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης των επόμενων χρόνο εμείς ως ε, ε, οργανισμός υποστηρίζουμε όσο γίνεται το ίδιο το Συμβούλιο μέχρι ότου, ε, μάλλον οποιοδήποτε σχήμα και αν έχει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω κάποιες από τις ε, προκλήσεις. Ε, καταρχήν υπάρχει ανάγκη το Συμβούλιο να είναι σε θέση να αναφέρεται πιο σωστά και πιο συνολικά σε αυτό που, ε, αποτελ... που αναφέρουμε ως χρόνιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο έχει επιδείξει δυνατότητα, ικανότητα να αντιμετωπίσει κάποιες επίγουσες καταστάσεις σε... με ειδικές συνόδους, αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των των ενημερώσεων, ο ύπατος αρμοστής αναφέρθηκε σε πολλές χώρες από όλες τις περιοχές του κόσμου όπου υπάρχουν δυσκολίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό βασίζεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ξεφύγει με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν υπάρχει κανένας παράδεισος για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί της γης. Αυτό μας βοηθά να βρούμε τρόπους και μας θυμίζει διαρκώς ότι υπάρχουν διαρκώς προβλήματα το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο διαφόρων πλαίσιων, είτε στο πλαίσιο των γενικών συζητήσεων ε, κατά τη διάρκεια των ειδικών συνόδων, εξετάζοντα ε, ε, εκθέσει των ειδικών εισηγητών, είτε ασχολούμενοι με ειδικού εισηγητέ για συγκεκριμένε χώρε, είτε ασχολούμενοι με το UPR. Όσον αφορά την διαδικασία UPR, το εργαλείο τα, τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το Συμβουλίο είναι τα ίδια με αυτά που είχε και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά δεδομένου του υψηλού επίπεδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του στάτου του και του προφίλ του, το Συμβούλιο είναι πάντοτε, έχει πάντοτε πολιτικό χαρακτήρα. Υπάρχει χώρο για βελτίωση προ αυτό το θέμα και θα ήθελα να ε, επενέσω, να εγκομιάσω τι προσπάθειε του Προέδρου του Συμβουλίου και του ίδιου του Συμβουλίου, ώστε να συμμετέχουν όλοι, όλοι τα μέλη του σε αξιοπρεπή συζήτηση. Αυτό που είναι Σημαντικό είναι να προσαρμοστούμε στο μόνιμο επίπεδο πολιτικού χαρακτήρα και να βρούμε μια λειτουργική διαδικασία ώστε το Συμβούλιο να είναι ένα πολύ ευέλικτο σώμα το οποίο να είναι σε θέση να συζητήσει κάθε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, η ευαλιξία στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα θα μπορούσε να επεκταθεί. Η, είπατε η αρμοστής ε, πολλές φορές αναφέρθηκε στις ειδικές ε, ε, ειδικέ συνεδριάσει κατά τη διάρκεια των συνόδων καθώ και δηλώσει του Συμβουλίου προ τον τύπο. Ω προ αυτό υπάρχει χώρο για δημιουργικότητα ώστε να έχει το Συμβούλιο μια, ένα ευρύτερο φάσμα μηχανισμών που ασχολείται, θα ασχολείται με διάφορε προβληματικέ καταστάσει. Εμεί θα πρέπει να προβλέψουμε το Συμβούλιο, να φανταστούμε μάλλον το Συμβούλιο με ευρύ και πιο καινοτόμο τρόπο. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο πώ είναι ένα παραδοσιακό σώμα του ΟΗΕ που συνεδριάζει ε, πολλέ φορέ το χρόνο στην όμορφη Γενέβη, μετά ακολουθώντας ένα άκαμπτο και περίπλοκο πλαίσιο, θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα από αυτά. Θα πρέπει να είναι ένα φόρουμ όπου θα, φόρουμ, όπου θα γίνονται ε, η ολομέλεια της Συνόδου, θα γίνονται οι διάφορες παράλληλες συνεδριάσεις, εκατοντάδες συμμετέχοντες, ε, εκπρόσωποι του τύπου και της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούν να συμμετέχουν. Τρίτον, η απαραίτητη ευελιξία θα μπορούσε να σχετίζεται με διάφορε ε, πτυχέ τη εργασία του Συμβουλίου. Είναι εξαιρετικό να οργανώνονται πάνελ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο λειτουργία. Σαφώ είναι μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, αλλά υπάρχει χώρο για να διαβεβαιώσουμε ότι η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων και άλλων ε, οργανισμών ή ε, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσε να είναι ε, ε, μεγαλύτερη. Εγώ προσβλέπω στις δικές σας προτάσεις ε, σχετικά με αυτό το θέμα σήμερα. Η δική σας εμπειρία σίγουρα θα μας είναι πολύτιμη. Η σημερινή επέκταση των πάνελ, 6 τον επόμενο Μάρτιο για την Σύνοδο, για παράδειγμα, θα μα οδηγήσει σε ένα τέταρτο στοιχείο, δηλαδή πώ θα ασχοληθούμε με την παραδοσιακή δραστηριότητα του Συμβουλίου ω σώμα του ΟΗΕ, δηλαδή τι γενικέ συζητήσει που είναι χαρακτηριστικέ οποιασδήποτε συνεδρίαση του ΟΗΕ και που παρέχονται ευκαιρίε για όλα τα μέλη και τους, τα κράτη παρατηρητέ να θέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η κοινωνία των πολιτών έχει επίση τη δυνατότητα να, να συμβάλλει σε τέτοιε συζητήσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο είναι χρονοβόρο και επαναληπτικό. καθώς και εξαιρετικά ευρύ στη φύση του. Γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα επαναδιοργανώσουμε το πρόγραμμα εργασίας μας. Μια άλλη σκέψη αφορά το μέλλον του UPR, όπου θα πρέπει σαφώ ε, ο εστιασμός της προσοχής μας να δοθεί στη συνέχεια που θα δοθεί στις συστάσεις. Αυτή τη στιγμή όλες οι συστάσεις που γίνονται από τους συμμετέχοντες στην ε, έκθεση ε, συγκεντρώνονται από τις εκθέσεις και, ε, από την UPR μάλλον και γίνονται, ε, γίνεται η εξέταση αυτών. Έχουμε 23.040 συστάσεις αυτή τη στιγμή. Πώς θα καταφέρουμε να δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά. Σαφώς και είναι πρόκληση για όλους. Ε, θα πρέπει να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς για να συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μέσα σε ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει στον εντοπισμό προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας η ιδέα ενός καθαριστικού κέντρου ε, ετέθη πριν από καιρό και μήπω. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το θέμα. Θα σήμαινε ότι θα γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο ε, ε, συνεδριάσεις με εκπροσώπους της υπηρεσίας, με ειδικευμένε υπηρεσίες, εκπροσώπους του ΟΗΕ, άλλες κυβερνητικέ οργανώσεις και ΜΚΟ. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τη μορφή των συστάσεων UPR αφού αυτή τη στιγμή η μορφή μιας ε, ενός τέτοιου εγγράφου του ΟΗΕ συμπεριλαμβάνει 120 διμερείς συστάσεις χωρίς ξεκάθαρη προσύστημα για να δούμε αν θα υποστηριχτούν ή αν θα απορριφθούν. Αυτό μας ανησυχεί. Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω τώρα. Πραγματικά ε, θα πρέπει να γίνει μια δυναμική ανταλλαγή απόψεων στην υποεπιτροπή σας. Είμαι έτοιμος να ακούσω τις απόψεις σας και σίγουρα όλα αυτά τα θέματα θα επανεξεταστούν ώστε να εξευρεθεί ε, μια μέθοδος εργασίας και ρυθμίσεις ε, και να γίνουν και οι απαντήστοιχες συστάσεις προς το Συμβούλιο. Ό,τι και να αποφασιστεί τελικά το 2000, μέχρι το 2011 θεωρώ πως είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση και να εστιάσουμε την προσοχή στην προσαρμογή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών και των δυνητικών θυμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τίστουνε για αυτή την πολύ συγκεκριμένη και ενδιαφέρουσα δήλωση για τα όσα κάνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος ε, της ε, Διεθνούς Αμνηστίας, ο κ. David Nichols. Επίσης, ο κύριος Αμασόλτ, που είναι, που είναι Πρόεδρο τη ε, Αρμόδιας Επιτροπή σα δίνω το λόγο για να σχολιάσετε τι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω στα σχόλια στα οποία προέβη ο Πρέσβη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν ήταν ένα από του ισχυρότερου υποστηρικτές ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι στιγμή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, ιδιαίτερα με την έκθεση Αντρικέν νωρίτερα φέτο και εθώς και τι πολυάριθμε αντιπροσωπείε που στέλνει το Κοινοβούλιο στην Γενέβη συνέβη. Σαφές είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη μέχρι και το τέλος της ε, φάσης ε, αναθεώρησης. Εμείς έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις και τις έχουμε υποβάλει στην Ένωση και στον πρέσβη όταν θα ε, χρειαστεί να γίνει η αναθεώρηση. Το πρώτο σημείο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουμε αποτελεσματικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί μόλι ολοκληρώθηκε η πρώτη γνήσια, ε, το πρώτο γνήσιο έτος εργασίας του Συμβουλίου, γιατί τα πρώτα δύο χρόνια δαπανήθηκαν ε, σε εσωτερική ρυθμίσει, ε, λειτουργία του θεσμικού αυτού οργάνου και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Συμβούλιο. Και υπάρχει ένας φόβος ότι αν στραφούμε και πάλι στην δομή και στις διαδικασίες θα αφαιρέσουμε την προσοχή από ε, την ε, πρακτική δουλειά του Συμβουλίου και γι' αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερα τη δήλωση που κάνατε ότι, Πρόεδρε, ότι δεν θα αποσπαστεί η προσοχή από την καθημερινή εργασία του Συμβουλίου λόγω της αναθεώρησης. Τώρα, αξιολόγηση της εφαρμογής των όσων ήδη έχουν συμφωνηθεί από το Συμβούλιο. Να μην ανοιχτεί δηλαδή και πάλι το πακέτο, της, ε, το διαδικαστικό, το λειτουργικό. Ορισμένοι μιλούν ότι, το, λένε ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα αποδώσει όσον αφορά την εντολή του. Ας πούμε, το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό αναφέρθηκε και από τον ε, Συμβούλιο στην, ε, ε, στο γραφείο της ΣΥΠΑ του Αρμοστή. Αυτό όμως δεν οφείλεται στην εντολή των ίδια, αλλά οφείλεται στο ότι δεν έχει ακόμα πλήρως εφαρμοστεί η εντολή. Όπως είδαμε εμείς από την ε, μερική αυτή εμπειρία, ιδιαίτερα μέσω της ε, φάσης, κατά τη διάρκεια μάλλον της φάσης οικοδόμησης των θεσμικών ε, διαδικασιών, θεωρήσαμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μέσω άτυπων συζητήσεων και όχι μέσω των επισήμων ομάδων εργασίας. Οι συζητήσεις ε, οδήγησαν στη δημιουργία δύο πακέτων θεσμικών και ήταν πολύ άκαμπτο αυτό. Οι θέσει των ομάδων φάνηκε να, επηρεά... να κυριαρχούν στις συζητήσει και αν ε, η διαδικασία λειτουργίας που τώρα έχει θεσπιστεί θέλουμε να βελτιωθεί, θα πρέπει να γίνει μια πραγματική ειλικρινή συζήτηση πέρα από τους περιορισμού των θέσεων των ομάδων, των διαφόρων ομάδων χωρών και την κυριαρχία των ε, μεγάλων χωρών σε αυτές τις ομάδες. Το Συμβούλιο και τα μέλη του δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της ε, αναθεώρησης για να προβούν σε βελτιώσεις στη λειτουργία του Συμβουλίου. Είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη ανάγκη για βελτίωση και στη λειτουργία του Συμβουλίου αφορά την συμπεριφορά των ίδιων των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις μεθόδου εργασίας τους. Υπάρχει σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα στη εργασία του Συμβουλίου, ενώ Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πολλά κράτη. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αντιπαράθεση που χαρακτηρίζει πολλές από τις εργασίες του Συμβουλίου. Επίσης, πολλές φορές ε, ισχυρά μέλη ε, υπαγορεύουν τις θέσεις των ομάδων χωρών. Το να αλλάξει η νοοτροπία λειτουργίας ε, δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί μέσω αυτή τη αναθεώρηση. Όμω θα πρέπει να προτείνει αυτή η αναθεώρηση πρακτικά μέτρα για να βοηθηθεί για να αλλάξουν οι πρακτικές μέθοδοι εργασίας. Όσον αφορά ε, μεθόδους εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωση εντός της, ε, του Συμβουλίου, έχουν υπάρξει βελτιώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την ευελιξία την κατανομή του φόρτου και την ε, πρόσβαση προς άλλες περιοχές, άλλες περιφέρειες. Εντό τη Ένωση θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στι περιπτώσει όπου είναι δύσκολο ή αδύνατο ε, να φτάσει σε συνένεση η Ένωση. Πολύ συχνά οι δυσκολίε συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν σε συνενεση η ενωση πολυ συχνα οι δυσκολιε συνενεση ευρωπαικη ενωση οδηγουν σε αδρανεια την Ένωση. Σε αυτέ τι ε, περιστάσει, το να επιτευχθεί κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον τον βασικό στόχο παρά το να επιτευχθεί μια ρεαλιστική συμφωνία λειτουργική με τι άλλε χώρε και τι άλλε περιφέρειες. Και αυτό το είδαμε χαρακτηριστικά ε, στην εργασία για την έκθεση Goldstone όπου η συζήτηση τη Ένωση για τη σύσταση την ουσία κυριάρχησε στη συζήτηση όχι μόνο στην πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου αλλά και στην ειδική σύνοδο αλλά και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης την περασμένη εβδομάδα και στη, και στη σχετική συζήτηση. Πολλά από αυτά που εμείς θεωρούμε ως βασικές προαπαιτήσεις για την εργασία του Συμβουλίου είναι μεγαλύτερη προσοχή σε καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν οφθαλμοφανείς και συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ε, προεδρικές δηλώσεις και προεδρικές ε, ανακοινωθέντα τύπου, καλύτερη συνεργασία των κρατών με τις ειδικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που καθεκαθιστούν ευκολότερο το, τις, για τις ΜΚΟ που δεν εκπροσωπούνται στην Γενέβη να απευθύνονται στο Συμβούλιο. Η ΜΚΟ θα πρέπει επίσης να είναι πλήρη μέλη της αναθεώρησης, να συμμετέχουν μάλλον πλήρως στην αναθεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει μεγάλη προσήλωση στην διαδικασία UPR, έχει εκπονήσει εκθέσεις και ίδια ε, και όπως ήδη υπόθηκε, το κλειδί για την ε, λειτουργία της διαδικασίας UPR είναι ακριβώς πώς θα δοθεί συνέχεια σε αυτές τις διαδικασίες. Η σημερινή πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεσχιστεί και να ενισχυθεί με συστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά σημεία για την συνέχεια που δίνεται σε αυτές τις εκθέσεις. Να δούμε δηλαδή, να δει και το Κοινοβούλιο πώς μπορεί καλύτερα να εντάξει τις συστάσεις των UPR στα δικά του ψηφίσματα και εκθέσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας, τις επικοδομητικές. Κυρία Αμαρσόλντε θα πάρει το λόγο αυτή τη στιγμή, εξ εξονόματος του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, εξαιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ και έτσι μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τη, δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να, ευχα... να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία ε... της παρουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου, τον κύριο Βαν Μέβεν και μέσω του κύριου Τίστονέ ε, να στηρίξω την εργασία της ΥΠΑ του αρμοστού και της υπηρεσίας της. Ε, όταν σας μίλησα για τις δικές μας προτεραιότητες, ανέφερα ότι η, το Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια από αυτές μας τις προτεραιότητες. Εμείς θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε ότι θα ε, εκπληρώσει την εντολή του το Συμβούλιο αυτό. Ε, ε, όπως έχουν παρατηρήσει και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, υπήρξαν πολλά επιτεύγματα από πλευρά του Συμβουλίου, αλλά ακόμα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Θα ήθελα να πω δύο σύντομα λόγια για τη δουλειά που κάναμε στις δύο συνόδους που έγιναν κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και να προβώ μετά σε δύο γενικότερα σχόλια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καθώς προετοιμαζόμασταν για την τακτική σύνοδο του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντόπισε ως προτεραιότητα τη συνέχιση των εντολών και των ειδικών διαδικασιών για τη Σομαλία, την Καμπότζη και τον Μπουρούντι αυτό ε, επετεύχθη. Επιπλέον, η ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε ένα ψήφισμα που ζητά την απελευθέρωση της Άνιεν Σουκή στην Βυρμανία, Μιανμάρ και μετά από έντονες πιέσεις επετεύχθη η υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος ομόφωνα στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο. Αναφέρθηκε και διάφορα άλλα σημαντικά ψηφίσματα. Το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα ε, για την Ανδούρα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρωτοβουλία Αιγύπτου, ΟΗΕ, για την υιοθέτηση για ένα ψήφισμα για την ελευθεροτυπία και ελευθερία έκφρασης υποβλήθηκε και εκεί καλωσορίσαμε την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι προηγούμενες, οι προηγούμε, τα προηγούμενοι μηχανισμοί και μετά από διαπραγματεύσει επετέφθη ψήφισμα το οποίο μπορούσε να υποστηρίξει η Ένωση και ήταν σημαντικό να μην υποχωρήσουμε από τις θέσεις που είχαν θεσπιστεί κατά τη διάρκεια της ε, αναθεώρησης ΔΕΒΟΝ καθώς και της ενημέρωσης ε, και, μάλλον ε, της έκθεσης για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Επίσης, ε, ε, ε, γίνανε ψηφίσματα για τη φτώχεια και την ε, υγειονομική περίθαλψη Ε, η δικαστή Γκόλστον επίση ε, έβαλε το ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη καθώ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και εκεί ε, υποχρέωση όλων των μερών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο την, αρχή, ε, την αρχή της ε, λογοδοσίας καθώς και σημαντικές άλλες δεσμεύσεις αναλήφθησαν από τα μέρη καθώς και υποστηρίχθηκε η συνέχιση και η παρακολούθηση της κατάστασης. Εμείς ενεργά είχαμε επαφές με τις αντιπροσωπείες των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών και συνεργαστήκαμε με την Παλαιστινιακή αντιπροσωπεία για να αποτύχουμε ένα ψήφισμα στην Ειδική Σύνοδο ένα ψήφισμα το οποίο να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ως Ένωση, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Άλλο σημαντικό ήταν η ετήσια εκδήλωση για τα φύλλα που ήταν από τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες των νέων διαδικασιών του Συμβουλίου. Στο μέλλον η Ένωση θα δώσει βέβαια μεγάλη προτεραιότητα στην διαδικασία αναθεώρησης. Τώρα που υπάρχει απόφαση να αρχίσει αυτή του χρόνου σε ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο άρχισε και η ανάλυση μεταξύ μας του πώς θα γίνει αλλά ήδη και οι συνεννοήσεις με άλλους εταίρους για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε καλύτερα να οργανωθεί η μελέτη αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Συμβούλιο, για το μέλλον. Και τέλος, στις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου. Ξέρω ότι είναι θέμα που η υποεπιτροπή σας το προσέχει ιδιαίτερα. Τέσσερα θέματα, τέσσερα. Ένα, η Ένωση παραμένει φάση πρωταγωνιστής στον αγώνα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι σωστό. Μόνο έτσι το Συμβούλιο θα μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και πρέπει στο εξής να συνεχίσει να επιμένει στην ε, υποστήριξη της ανεξαρτησίας της υπάτης αρμοστίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συνεισφέρει και αυτή στην εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το γενικότερο θέμα που θα έπρεπε να θίξουμε εδώ είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα πρότυπα που καθόρισαν, που έχουν υποχρέωση μάλλον να σέβονται τα μέλη του ΟΗΕ. Δεύτερον, έχουν αυξηθεί οι προσπάθειές μας για αύξηση της συνεργασίας. Πριν από τη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου είχαμε οργανώσει δύο γύρους outreach, outreach για να μιλήσουμε για θέματα που προβλέπονταν από τις μελλοντικέ ημερήσιες διατάξεις μας αλλά και να εξηγήσουμε τις πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της Ένωσης. Και οι επαφές με άλλους εταίρους ήταν ιδιαίτερα έντονες για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είπατε και εσείς σήμερα, καμιά φορά ακούγονται κριτικές κατά της Ένωσης ότι στον ΟΗΕ αντιδρά πολύ μονολυθικά. Γνωρίζουμε και εμείς ότι πρέπει να αυξηθεί η ομαδική δυναμική της παρουσίας μας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα αποτελέσματα. Τα απαντήσαμε στις επικρίσεις που ακούστηκαν και προσπαθήσαμε τη συμμετοχή της Ένωσης να την κάνουμε στο εξής με περισσότερες φωνές γιατί καμιά φορά η πολυφωνία αλλά και η ομοφωνία είναι καλό αποτέλεσμα. Ο διαδραστικός διάλογος όπως λένε είναι νομίζω ένας τρόπος βελτίωσης της δυναμικής της λειτουργίας του Συμβουλίου. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι η Ένωση δεν συντονίζει θέσεις και δηλώσεις δεν συντονίζει. Τρίτον, τις διαδικαστικές συζητήσεις τις κάναμε πιο ενεργά και πιο διαδραστικά και αυτές. Στο, το Σεπτέμβριο ας πούμε η Ένωση παρενέβη για να υποστηρίξει τα δικαιώματα ορισμένων μήκη όμικρων. Τέλος, συμφωνώ ότι με τον κύριο Τιστονέ ότι ακόμα παραμένει πρόκληση η καινοτομία για μας και η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να μας δώσει το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος Συμβουλίου γιατί συνεχίζει το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για την για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στο βάθος της εθούσης θα έχετε δει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παρατηρητών. Είναι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αλγερίας, της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, αλλά και μια ομάδα βουδιστών μοναχών από την Βυρμανία που ήρθαν γιατί ανησυχούν ιδιαίτερα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Και αυτό είναι και θέμα που αφορά την και την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας τους. Αν μπορέσουμε θα τους δώσουμε το λόγο στο τέλος της συνεδρίασης. Αλλά πρώτα πρέπει να εξαντλήσουμε την μερίσια διάταξη και να οργανώσουμε και τη συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων. Κυρία Μπρέπολ, Νίλσεν, Γκόμε, Τάνοκ, Γουίτ και άλλο. Ζητάει κανεί άλλο το λόγο, ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Ο κύριο Χόουι, δεν τον είπα, τον είπα πριν. Ο κυρία Μπρέπολ αρχίζει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο μας χορήγησαν τις πληροφορίες τους. Καθώς και για την κριτική που άσκησαν, την αυτοκριτική μάλλον. Η κριτική αυτή βέβαια δεν υποβιβάζει το ρόλο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απλώς εννοεί ότι ο οι ίδιες οι χώρες καμιά φορά ε, μέλη παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως τίθεται το ερώτημα του τρόπου με τον οποίο μπαίνουν οι χώρες αυτές στο Συμβούλιο. Αν δείτε το κείμενο που πρότεινε το Πακιστάν, θα διαπιστώσετε ότι αφορά προώθηση θρησκευτικού μίσους, μυσαλλοδοξίας. Τι αξιοπιστία προσδίδει αυτό στο Συμβούλιο. Καμία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία της έκθεσης Goldstone. Εγκρίθηκε με πολύ δύσκολα, με μεγάλη δυσκολία και αν δει κανείς πόσοι χώρες μέλη συμπεριφέρθηκαν θα διαπιστώσει επίσης ότι τώρα που θα υποβληθεί έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα υπάρξουν απορίες και ερωτήματα είναι σημαντική βέβαια η έκθεση για να μην υπάρχει ατιμορρησία και να υπάρχει αντίθετα λογοδοσία. Να θεωρούνται υπεύθυνε ορισμένες χώρες για ό,τι έχουν διαπράξει. Αλλά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΣΑΔ, δεν θα μπορέσει μάλλον να αλλάξει τα πράγματα και να επιβάλλει να γίνει κάτι για να τιμωρηθούν οι υπέτειοι. Άρα εδώ φαίνεται ότι στο Συμβούλιο διαφαίνεται ότι υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες, δηλαδή μερικές χώρες του, μέλη του είναι κατά των δυτικών αξιών και άλλες απλώς διαφωνούν και θεωρητικά με τους στόχους του. Τι εγγυήσεις μπορούμε να έχουμε λοιπόν ότι θα γίνει μια αντικειμενική έρευνα του τι έγινε κατά τις επιθέσεις στη Λουρίδα της Γάζης. Ευχαριστούμε κυρία Μπρέπολς. Γκόμες. Ευχαριστώ και εγώ τους παρεμβαίνοντες και εγώ θα ακολουθήσω την Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι με κοιτούσατε και είχα βγάλει ήδη τα ακουστικά μου. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, και εσείς είσαστε στο κατάλογο των ομιλητών, αλλά προσπαθούμε να καταρχήν να, εναλλάξουμε τους εκπροσώπους διαφόρων πολιτικών ομάδων. Γι' αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα την κυρία Γκόμες να παρέμβει. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι ε, πριν 20 ε, χρόνια ήμουνα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ε, καταρτήσουμε ένα ψήφισμα για την Ρουμανία και την Μιανμάρ. Ευτυχώς όμως ε, η Ρουμανία ακολούθησε πορεία μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου ε, αλλά στο μιαμάρι η κατάσταση δεν είναι καλύτερη μετά από 20 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να ε, υπερψηφίσουμε το ψήφισμα για τη οάν Σαν Σουσί. Όταν έφυγα από την ε, ε, Επιτροπή το 1994 είχαμε πολλές αμφιβολίες για τις αλλαγές στο Συμβούλιο και ε, αυτά τα οποία έγιναν ε, επιβεβαίωσαν τις δισταγμούς μας διότι ναι ε, ε, πρέπει να διατηρήσουμε την, τους δύο οργανισμούς αλλά και ε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι πολιτικοποιημένη. Είναι πολιτική και πολύ σωστά, διότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο της πολιτικής και βεβαίως οι διαφορές είναι ότι τώρα οι παραβιαστές ε, έχουν αποφασίσει να υπησέλθουν ε, και να παρεμβάλλουν σε όλους τους οργανισμούς και στα μέσα που έχουμε είχαμε παλιά δυστυχώς δύο μέτρα και δύο σταθμά τα οποία ούτως ή άλλως ε, δεν είναι προς όφελόν μας, και είμαστε ε, ε, παραλυμένοι διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και όπως ελέγχθη από τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας ο οποίος ε, έχει αναφέρει το παράδειγμα ε, πρέπει να προχωρήσουμε αλλά ε, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις νομίζω ότι οι δύο αλληλεπιδράσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και του ομολόγου της Επιτροπής είναι χρήσιμη τότε και εγώ ήμουν εκπρόσωπος της Επιτροπής και δεν μπορώ να παρέμβω, αλλά πιστεύω ότι όσο νωρίτερα εμπλακούμε τόσο περισσότερο θα αποδώσουμε. και σιγά σιγά οι κυβερνήσεις και ακόμη και οι διπλωμάτες θα μπορέσουν να αντιληφθούν τα προσόντα της, του καθεστώτος αυτού. Θα ήθελα επίσης να, σα, να ρωτήσω εάν υπάρχει μία βελτίωση, αν υπάρχει κάποια βελτίωση τώρα που έχουμε τη δίκηση ο Ομπάμα, με την οποία υποτίθεται ότι έχουμε περισσότερα κοινά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα από ό,τι είχαμε παραδείγματο χάρη με την διοίκηση Μπούς. Και το τρίτο μου ερώτημα είναι το εξής δεν είναι κριτήριο ότι πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο να χρησιμοποιήσουμε το Συμβούλιο και να κατανείμουμε τις ε, ευθύνες προς το Συμβούλιο ε, δεν θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να διερευνούμε περισσότερο τα πράγματα με πιο καινοτόμους μεθόδους. Ε, είχαμε συζητήσει για την Ερυθρέα παραδείγματος χάρη πρόσφατα και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ εννοούμε και από πλευράς οικονομικής, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι ε, υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, αυτό επίσης είναι κάτι που μπορεί ε, να γίνει στο επίπεδο του Συμβουλίου. Τώρα, τι γίνεται στη Ζιμπάμπουε. Άπαξ και ο ειδικό εισηγητή ε, εξεδιώχθη χωρίς καν να μπορέσει να καταρτήσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ασυνήθιστα συμφωνώ σχεδόν με όλα που είπε η Άννα Γκόμες, το οποίο είναι ανησυχητικό διότι και εγώ στην αρχή ήλπιζα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 αξιοπιστία είναι ίσως λίγο περιορισμένη όταν μιλάμε για την Σαουδική Αραβία η οποία ε, θεωρεί ότι τα οικονομικά εγκλήματα αξίζουν την ποινή θανάτου στο Πακιστάν. Δηλαδή αναφέρουμε εδώ σε διάφορα μέλη τα οποία ε, είναι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο αυτό και όλοι επικεντρώνονται στο θέμα του Ισραήλ και ε, των Παλαιστινίων με 25 ε, φορές περισσότερα ψηφίσματα κατά του Ισραήλ πράγμα το οποίο δείχνει σαφώς μία μία τελείως μονομερή αντιμετώπιση. Επίσης δεν έχει αναφερθεί ότι είχαν ε, ε, σταλεί ε, πολλά πολλά Eh, eh, eh, Πολύ πύραυλοι κατά του Ισραήλ και τελικώς ε, όπου η αμερομηψία του Συμβουλίου Αυτούνου δεν είναι αποδεδειγμένη δηλαδή αυτό δυστυχώς δείχνει σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στους Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ και, και εγώ διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι στην Επιτροπή υπάρχει ομοφωνία και ότι εσείς συμφωνείτε με την κυρία Γκόμες. Ε, η κυρία Κίνετσεν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή της συνεδριάσεως αναφερθήκατε στην επέτειο της ε, καταρρύψεως του τείχους στη Γερμανία ε, αλλά βρισκόμουν στην ε, Δυτική Όχθη πρόσφατα και όπου δεν καταστρέφουν τα τείχη αλλά σκέφτονται σκέφτονται να δημιουργήσουν ένα τείχος που θα αποκόπτει ακόμη και τους γεωργούς από τα χωράφια τους και τα παιδιά από το σχολείο τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που πήγα σε αυτή την περιοχή και διαπίστωσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ άτομα τα οποία εξεδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν ζήσει 33 χρόνια στα, σπίτι, σπίτια αυτά τη νύχτα εξεδιώχθηκαν και την επομένη το πρωί αντικαταστάθηκαν με κατοίκους ε, απίκους Ισρα... Ε, ε, Ισραηλινούς βέβαια ξέρετε ότι η περιοχή αυτή έχει πληγεί διαμέσου των ετών από διάφορες κατοχές Βρετανική, Οθωμανική ε, τώρα Ισραηλινοί και τέτοιες ε, περιστάσεις υπάρχουν πολλές αφού εξεδιώθηκαν, εξεδιώχθηκε ε, κάποιος από την ε, Δυτική Ιερουσαλήμ το 48 με, στη συνέχεια εξεδιώχθη παρόλο που και άλλοι ε, είχαν μείνει σε αυτά τα σπίτια ε, δικαιωματικά από 33 ετών εξεδιώχθηκαν σε μία νύχτα είτε πρόκειται για ηλικιωμένους είτε για νέους. Θέλω λοιπόν εδώ να καταφερθώ κατά της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή και να σας πω ότι υπάρχει και το δικαίωμα ε, για ίδρευση που είναι επίσης ένα δικαίωμα όλων και η Διεθνής Αμνηστία ε, καταγγέλει την ε, κατοχή του, των υδατίνων πόρων από το Ισραήλ ε, εις βάρος των Παλαιστινίων και οι Ισραηλινοί καταναλώνουν 20, 20 φορές περισσότερο νερό από ότι οι Παλαιστίνοι στην περιοχή. Επίσης στη Γάζα όπου είναι αποκλεισμένο ένα εκατομμύριο άτομα μετά από έναν πόλεμο όπου υπάρχει ελάχιστο νερό μόνο 10% του νερού της Γάζας σέβεται ε, τις ε, διατάξεις και προδιαγραφές του ΠΟΗ, δηλαδή είναι πόσιμο και θέλω ε, να καταγγείλω την ατιμορρησία του κράτους του Ισραήλ που αποτελεί ένα παράδειγμα κάποιας δημοκρατίας στην περιοχή και πιστεύω ότι αυτή η ατιμορρησία ε, διακινδυνεύει τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και επιτρέπει σε δικτάτορες και σε χούντες να χαίρουν σε ορισμένες περιοχές ε, κάθε ευημερία και δεύτερον ε, μία ερώτηση που έχει ήδη τεθεί τι γίνεται με την έκθεση Γκόλσον τι συνέχεια πρόκειται να δοθεί στην έκθεση αυτή σας ευχαριστώ ευχαριστώ η κυρία Γκέτ Νίλσεν Εδώ μιλάμε με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ο κύριος Βαν Μέβεν προφανώς θα αναφερθεί στη διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, ε, εάν θέλει. Έχω όμως και άλλα ονόματα στον καταλογά μου, ο κύριος Χάουιτ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Πρέσβη. Ευπρόσδεκτη ευκαιρία να συνομιλήσουμε άμεσα. Εγώ ήμουν μόνιμος μέλος ε, της αποστολής μας ε, στη Γενέβη. Είχα αυτό το προνόμιο. Ήμουν ε, μέσα στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίξαμε ελπίζω έναν επικοδομητικό ρόλο συνομιλώντας με τους πρέσβους μας εκεί και ε, βοηθώντας τους να λάβουν υπόψη τα τις θέσεις μας, αλλά και αποτελώντας μέλος αυτής της ευρωπαϊκής ε, ε, πλευράς της, Ευρωπα... της ευρωπαϊκής φωνής εκεί, που ελπίζουμε ότι ακούγεται. Η στόχοι του Κόφεναν, όταν συμφωνήθηκε η πρώτη αναθεώρηση, Ελπίζε ότι θα ήμασταν πιο το Συμβούλιο θα ήταν πιο αντικειμενικό, λιγότερο πολιτικού χαρακτήρα, Όλοι το ελπίζαμε αυτό και θα πρέπει να πω ότι απογοητευθήκαμε. Δεν σας επικρίνουμε εσά και τη θέση σας, αλλά νομίζω πως ε, είναι δίκαιο όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ε, όθηση της υπόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλες αυτές οι προσδοκίες δεν υλοποιήθηκαν στο βαθμό που ελπίζαμε. Είναι σαφές και παράδειγμα ότι τα παλαιστινιακά εδάφη πραγματικά έχουν επηρεάσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε έντονα αισθήματα περί αυτού, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέχρι και την τελευταία εβδομάδα που προσπαθήκαμε να προσπαθήσαμε να βρούμε λύσει σε αυτό το θέμα, είναι δυσανάλογη η επίπτωση αυτών όλων στι, υπόλοιπε υποθέσει. υποθέσεις. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μέση Ανατολή και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά σίγουρα και εγώ το έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους και με την Σουηδική Προεδρία με την οποία έχουμε εξαιρετικές θέσεις, ε, σχέσεις, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει έναν ευρύ ρόλο για να βρεθεί μια γνήσια θέση για τα παλαιστινικά εδάφη που να είναι ισορροπημένη, θα λάβει, βάλει, βάνει υπόψη όλα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε εδώ, να βοηθήσουμε, θα πρέπει αυτό να το κάνουμε και θα μας ενδιαφέρει να μας απαντήσετε σε αυτό. Η Προεδρία έχει καταστήσει σαφές ότι ορισμένα από τα πράγματα που ήταν ψηφίσματα του Κοινοβουλίου ήταν ε, πλήρη, σε πλήρη συμφωνία με την Προεδρία για το κατά πόσο θέλουμε, μάλλον πώς θέλουμε να είναι το Συμβούλιο σε σχέση με την οργάνωσή του και τη λειτουργία του. Σίγουρα θέλουμε να προστατεύσουμε τις ειδικέ διαδικασίες και την ανεξαρτησία της ΥΠΑ του αρμοστού και να βελτιώσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτά είναι πράγματα που νομίζω θα ενδιαφέρουν όλους όσους ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι ακόμα είναι ότι στην έκθεσή μας εξετάσαμε και θα πρέπει να τα πούμε ένα θέμα είναι ότι στις εκλογές στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι χώρες που θέλουν να είναι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν ανοιχτή πρόσκληση στις ειδικέ διαδικασίε. Αυτό είναι κάτι, είναι η γραμμή που υποστηρίζει το Κοινοβούλιο και νομίζω πως δεν είναι άδικο αίτημα για κάποιον που θέλει να μπει στη λέσχη. Ε, επίσης, ε, όταν οι υποψήφιες χώρες ε, ε, θέλουν να εκλογούν στο Συμβούλιο, κάνουν κάποιες δηλώσεις. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί και ένα βαθμό λογοδοσίας για τα όσα... Κάπου μάλλον θα, γίνεται, θα πρέπει να γίνεται και η λογοδοσία για τις δηλώσεις αυτές και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. και για το πώς μπορούμε να το σκεφτούμε. Υπήρχαν πολύ ψηλέ προσδοκίες ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στα θέματα της υποτορμοστή ε, και τελικά από ό,τι κατάλαβα έχει υπάρξει γνήσι πρόοδος, ε, έχει υπάρξει συμβολή τονίζοντας κάποιες τις κριτικές, ε, τις επικρίσεις και τα σκληρία ερωτήματα, καλωσορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το UPR, αλλά υπάρχουν και κάποιες παράπλευρα, κάποια παράπλευρα προβλήματα, θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική. Επίσης υπόθηκε ότι αν δεν έχουμε μία φωνή δεν δίνουμε καλό παράδειγμα στις άλλες περιφερειακές ομάδες χωρών και εκπρόσωπο της ΜΚΟ εδώ μας είπε ότι ορισμένε φορές μας έχει βοηθήσει να συντονίσουμε τι θέσει μα. Δεν το λέω αυτό επικρίνοντα του Σουηδού συναδέλφου, αλλά είναι μια δυναμική που όλοι αντιμετωπίζουν, όλε οι προεδρίε αντιμετωπίζουν. Η μεγαλύτερη απειλή που πρέπει να του ανησυχεί είναι ότι μπορεί να υπάρξει διαφωνία ανάμεσα στα μέλη τη Ένωση. Και είναι λυπηρό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά ξέρω ότι η πίεση ασκείται στη Γενέβη για να υπάρχει διχόνοια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό η δικοί μας πρέσβεις να μην ακολουθούν αυτή την ε, πορεία. Να μην ανησυχούν για τις μικρές αδιαφορές απόψεις. Είμαστε, έχουμε ασκήσει τέτοιου είδους επικρίσεις και προς την Προεδρία και βλέπουμε ε, να μην το πω μόνο στην, να το πω στην Σουηδό ε, συνάδελφο, στη Σουηδή συνάδελφο, και μάλιστα ήμουν και στη Στοκχόλμη για να παρακολουθήσω τη διάσκεψη της δικής σας προεδρίας. Εδώ δεν μιλάμε για μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μιλάμε για τις μεμονωμένες χώρες που να είναι προετοιμασμένες να ε, συνενέσουν και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση. Είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ και που ήταν πολύτιμη δική σας παρουσία εδώ σήμερα κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Χάουιτ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαν και στην κυρία Αμαρσέτ. Πριν όμως δώσω το λόγο τελικά στον πρέσβη, πριν απαντήσει δηλαδή, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση. Έγινε λόγος για τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, ο οποίος επισκέφθηκε τη Ζιμπάμπουε και τα συμπεράσματά του ήταν αρκετά ανησυχητικά ότι υπάρχει νέο κύμα πολιτικής βίας στη χώρα αυτή. Ο κύριος Νόβακ παρατήρησα είπε ότι ίσως θα έπρεπε να επιτευχθεί κάποια γενική συμφωνία για το σεβασμό των διαδικασιών, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Το θέμα είναι σοβαρό και δεν περιορίζεται στη χώρα εκείνη. Σε πολλές χώρες σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα έπρεπε αυτό το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κάνει κάτι. Κύριος Βαν Μόλτερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προηγούμενους ομιλητές για όσα μας είπαν το απόγευμα και που θα μας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τη συνέχεια των εργασιών μας στη Γενέβη. Ήθελα να προσθέσω ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κάτι το πολύ καινούριο. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να επεξεργαστούμε τη λεγόμενη θεσμική δέσμη και γι' αυτό το Συμβούλιο Τώρα αρχίζει την ουσιώδη εργασία του, εδώ και με το ζόρι ένα χρόνο. Το να κρίνουμε λοιπόν ήδη από τώρα τα πεπραγμένα του είναι νομίζω κάτι πρόωρο. Δεν λέω βέβαια ότι μέχρι τώρα έχει σημειώσει καμία τεράστια επιτυχία. Πρέπει όμως να θυμάστε όπως είπε και ο διπλανός μου μιλητής ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση των διεθνών σχέσεων όπου η πολυπλευρικότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί αλλά ο κόσμος δεν μπορούμε παρά να δούμε ότι έχει αλλάξει και, και όσοι κυριαρχούσαν στο παρελθόν αυτή τη στιγμή μερικοί τουλάχιστον είναι βρίσκονται σε αμυντική θέση. Βέβαια δεν έχω καμία απλή απάντηση για όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό που ξέρω ότι χρειάζεται είναι να υπάρχει θέληση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη φαίνεται να συμμετάσχει στη λειτουργία του Συμβουλίου και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαιτέρως και για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών όπως και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται. Το Συμβούλιο είναι αυτό που θα ήθελαν να είναι τα μέλη του. Λειτουργεί περισσότερο ή λιγότερο καλά ανάλογα με το τι θεωρούν προτεραιότητα οι χώρες μέλη του στη διεθνή πολιτική. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο πολιτικό, γιατί είναι πολιτικό κυρίως όργανο τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εξόχως πολιτικό θέμα. Ακούστηκαν, ακούστηκε πολύ, έγινε πολλής λόγος το απόγευμα για την έκθεση Goldstone τη Μέση Ανατολή και θέλω να σας πω ότι οι διαφωνίες που ακούστηκαν εδώ μέσα αντικατοπτρίζονται ακριβώς σχεδόν και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η μόνη λύση θα ήταν να γίνει μία αντικειμενική εξέταση της έκθεσης από όλους τους ενδιαφερόμενους. Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης ζητάει από τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς να διεξαγάγουν μία ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα για τη Γάζα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ουσιώδες όντως για την αναθεώρηση τώρα. Νομίζω ότι είναι και αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Και το είπαν και οι προηγούμενοι. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη συνήθη δραστηριότητα του Συμβουλίου. Θα τη συνεχίσουμε και την κανονική του δραστηριότητα. Αλλά θα υπάρξει και αυτή η αναθεώρηση με στόχο όχι να ξαναρχίσουν όλα από την αρχή, να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του, ώστε να μπορεί το Συμβούλιο πιο εύκολα, πιο αποτελεσματικά να ανταποκρίνεται στους στόχους του. Μιλήσατε και για τη Ζιμπάμπουε και αν μου επιτρέπετε, επ' αυτού θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντίσου του Συμβουλίου μας, που είναι πιο ειδικό από μένα για αυτό το θέμα. Αν μου το επιτρέπετε βέβαια. Ευχαριστώ σας το επιτρέπουμε. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente du, du, du sous-comité. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι η οργάνωση κατάρτισης ενός ε, ειδικού εισηγητή για οποιαδήποτε περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ειδικέ διαδικασίες μέσω μιας επιτροπής η οποία επιλαμβάνεται του θέματος και στη συνέχεια θα μας υποδείξει διάφορα πράγματα, δηλαδή ε, το γεγονός ότι ήδη ε, πέρασε μία νύχτα σε ένα αεροδρόμιο χωρίς ε, να μπορέσει να, να ταξιδεύσει και ταξίδευσε μία μέρα μετά αλλά ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτή η επίσκεψη και γι' αυτό κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο ειδικό εισηγητής να μπορέσει να εκτελέσει την αποστολή του σαν αρμοστία αναλαμβάνουμε ε, το θέμα αυτό κάνουμε κάθε τι δυνατόν και θα ήθελα να σχολιάσω σχεδιάσω την πολιτικοποίηση του Συμβουλίου σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος προηγουμένως διότι η πολιτικοποίηση όπως ελέγχθηκε σήμερα θα παραμείνει πάντοτε ένα χαρακτηριστικό του Συμβουλίου, δηλαδή όσο πιο ψηλά φτάνει στην ιεραρχία των Ηνωμένων Εθνών, τόσο πιο πολυκοτικοποιημένο θα είναι και υπάρχουν θέματα σχετικά με τα βασανιστήρια ή με τη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια τα θέματα αυτά ποτέ δεν είναι ήρεμα πάντοτε υπάρχει πολιτικοποίηση οξία και το 2006 όταν έγινε μεταρρύθμιση είχαμε προτείνει να υπάρχει παγκοσμιοποίηση αλλά έκτοτε εγκαταλείψαμε την ιδέα διότι θεωρούμε ότι είτε είναι κάποιος πλήρες μέρος είτε απλώς παρατηρητής έχουν ε, ίσες ε, δυνατότητες και ίσα δικαιώματα και χρειαζόμαστε ε, να έχουμε μία ευελιξία κατά τρόπον ώστε να εξετάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού όπου κινδυνεύουν και εδώ αναφερόμαστε σε όλα τα κράτη του πλανήτη δηλαδή πουθενά τα δικαιώματα δεν την χάνουν πλήρης ε, πλήρου σεβασμού. Δεν πρέπει να ανοίγουμε όμως τα κουτιά της Πανδώρας, τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένω να μείνουν σφραγισμένα για πάντα. Ευχαριστώ κύριε Τριστουνέ και τώρα η κυρία Χάμερσκιόλτ σαν για την ολοκλήρωση του θέματος διότι έχουν υπάρξει διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις δηλαδή ιδίω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εμπλακούν περισσότερο στις εργασίες του Συμβουλίου επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως σημείωσα τις συγκεκριμένες προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στα ερωτήματα που μου τέθηκαν και θα ήθελα επίσης να σημειώσω την αλληλεπίδραση μεταξύ μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την επιρροή τους ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με διάφορους τρόπους. Είχα ενημερώσει την υποεπιτροπή σχετικά με ε, τις προθέσεις της Σουηδικής Προεδρίας για την εργασία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν από την τακτική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και είχα ακούσει τις ερωτήσεις που έθεσαν τότε τα μέλη, ε, οι ευρωβουλευτές. Τώρα ε, ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αλλά θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες όπου μέλη της υποεπιτροπής επισκέπτονται τη Γενέβη και τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί μπορούμε να διερευνήσουμε πώς να ε, συσφίξουμε τη συνεργασία μας. Ρωτήσατε σχετικά με τον ρόλο της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως ε, η η θέση αυτή σαν νέο μέλος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε. Έχουμε δει τις ε, επιπτώσεις, έχουμε πολύ στενή επαφή με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε νέους τρόπους να συνεργαστούμε σχετικά με την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου σε όλα τα θέματα. Μου ζητήσατε να σχολιάσω τις προοπτικές ε, εστιάσεως ε, σε κυβερνήσεις ε, οι οποίες υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβούλιο έχει έναν ρόλο με τρεις πτυχές καταρχήν να προσφέρουμε τεχνική βοήθεια που δεν έχει τόσο πολύ τονιστεί στη συζήτηση αλλά βοήθεια στις χώρες που θέλουν να βελτιώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένας βασικός μας στόχος. Δεύτερον, η υπεράσπιση του δικαιώματος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων εκπροσώπων να συμμετέχουν ε, στις εργασίες του Συμβουλίου. Υπάρχουν διάφορα τέτοια παραδείγματα και πρέπει να τα θυμόμαστε όσο προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Συμβουλίου και επιπλέον το Συμβούλιο όπως και η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας χώρος όπου όσοι θέλουν να αντιταχθούν στις ε, ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορέσουν να εισακουστούν. Άλλωστε το Συμβούλιο πρέπει επίσης να αναλάβει τις ευθύνες του και να ανταποκριθεί στις σοβαρές ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ε, αντιδράσει με διάφορους τρόπους. Ερωτήθηκα επίσης πόσο θα ήταν δυνατόν να υπάρξει συνένεση σε θέματα που αναφέρονται στη Μέση Ανατολή. Ε, είναι ένα βασικό θέμα και έχει στενή σχέση με την έκθεση Goldstone. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο έγινε και στην τακτική ε, ολομέλεια και στην έκτακτη ολομέλεια και διατυπώσαμε διάφορες ε, προτάσεις ε, χωρίς βέβαια να επιτύχουμε το στόχο μας τελικά αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να συνομιλήσει και να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους και το τελευταίο θέμα που ανέφερε ο κύριος Χάουιτ ε, στο, για το outreach, το οποίο δεν πρέπει να αποτελέσει το μοναδικό ρόλο της Προεδρίας. Υπάρχει κατανομή των βαρών όπου και άλλες οργανώσεις συμμετέχουν και γι' αυτό ε, υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να τονίσει ε, την, ε, ε, την ευρεία ποικιλία θεμάτων που πραγματεύεται η Προεδρία πέραν της τριμερούς Προεδρίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για τις προτάσεις τους και τις για τα σχόλιά τους και ιδίως ε, γιατί θα ε, επιτρέψουν να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Του χρόνου θα καταρτήσουμε μία έκθεση με συστάσεις σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, ενίσχυση και όλων των διαδικασιών κατά τρόπον ώστε το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα σε συγκεκριμένες χώρες. Θέλω όμως τώρα να ευχαριστήσω τον πρέσβη Βαν Μεύεν, τον κύριο Τριστουνέ, τον, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και την κυρία Χάμερ και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο θέμα της συνεδριάσεώς μας το οποίο είναι η ακρόαση σχετικά με θέματα ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια. Εδώ έχουμε τον κύριο Κούγκαν που είναι ο πρόεδρος και ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών για να μπορέσουν να καταλάβουν τις θέσεις τους οι νέοι εκπρόσωποι. Ευχαριστώ. No niin, kokous jatkuu. No niin, arvoisat valiokunnan jäsenet ja kaikki vieraat erityisesti. Λοιπόν, αγαπητά μέλη της Επιτροπής και αγαπητοί ε, κύριοι διπλωμάτες από τις βαλκανικές χώρες που παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση εδώ Έχουμε μία ακρόαση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια και θέλω να, να αναφέρω ιδιαίτερο στον κύριο Κούγκαν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τη σχέση με Αλβανία, Βοσνία και Ζεγοβίνη, Σερβία, Βρομβούνη και Κωσυφοπέδιο. αυτό θα κάνει και την εισαγωγή και θα μας ε, ε, ε, παρουσιάσει τη δικιά του εμπειρία. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι 14 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την έκθεσή της σχετικά με την με την πολιτική επεκτάσεως και εκεί θα βασιστούμε όσον αφορά τις ε, εκθέσεις προόδου για να δούμε ε, ποιες είναι οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί εις ε, τις πιθανές υποψήφιες χώρες τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στην Κροατία, στην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στην Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Θέλουμε εδώ να αναφερθούμε ιδιαιτέρως στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή και στην ε, διαδικασία ε, διαμεσολάβησης η οποία διεξάγεται αυτή την ε, εποχή. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Έντουαρτ Κούγκαν ο οποίος είναι ο επικεφαλής της αρμοδίας αντιπροσωπείας. Έχετε το λόγο κύριε Κούγκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, πρόσφατες εκθέσεις της ε, Επιτροπής για την κατάσταση που επικρατεί στα Δυτικά Βαλκάνια δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει, ότι δικαιολογείται ένα συγκρατημένος ενθουσιασμός για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις χώρες αυτές. Επίσης, διατυπώνουν μια έκκληση στις χώρες αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των κριτηρίων ένταξη, των ενταξιακών δηλαδή κριτηρίων, διότι ακόμη λείπουν πολλά για να συμπληρωθεί επιτυχώς αυτή η διαδικασία. Τα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης, μεταξύ των οποίων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των μειονοτήτων, είναι πολύ σημαντικός στόχος μεταξύ αυτών. Αυτό ακριβώς που συζητάμε και σήμερα δηλαδή. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει γίνει πρόοδος και στα προηγούμενα χρόνια αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα, με την κάθε χώρα. Και τις περισσότερες φορές οι προσδοκίες δεν ε, δικαιολογούνται από τα αποτελέσματα. Θα σας αναφέρω ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να συνεχίσουμε να τα προσέχουμε κατά την επόμενη περίοδο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Η συμφιλίωση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι το πρώτο μου θέμα. Θα έπρεπε να θεωρείται ως ένας από τους κύριους φραγμούς για τη διαδικασία σταθεροποίησης που άρχισε από το 2000. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες αναχώρα, γιατί νομίζω δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να αρχίσω με το δικαίωμα των προσφύγων και των, the priority is the promotion. και των εκτοπισμένων η πρόσβασή του σε βασικά δικαιώματα όπως στέγαση, παιδεία, υγεία, απασχόληση και κοινωνικές υπηρεσίες είναι προβληματική. Άλλο σημαντικό πρόβλημα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι η σοβαρή και υπεύθυνη τιμωρία των εγκλημάτων πολέμου και, και μετά η συμφιλίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα έχει δώσει κίνητρα στις χώρες αυτές για να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Νοτιοσλαβία. Και η εθνική τους δικαστική διαδικασία αντιμετώπισης των εγκληματιών είναι κάτι που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί στις χώρες αυτές. Σε πρόσφατα χρόνια οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έκαναν προσπάθειες για να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους σε διεθνή πρότυπα ως προς τις μειονότητες. Παρά κάποια πρόοδο που επιτεύχθηκε εκεί, η κατάσταση ακόμα δεν είναι ικανοποιητική. Ορίστε μερικά από τα προβλήματα που θέλω να Αυτά ήταν μάλλον μερικά από τα προβλήματα που θέλησα να σας αναφέρω, αλλά υπάρχει και το θέμα του μέλλοντος. Θα σας πω δηλαδή τώρα τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η κατάσταση των προσφύγων και των εσωτερικών εκτοπισμένων. Η βοήθεια των προσταθήματα. Πρόοδος της περιφερειακής συνεργασίας στο θέμα των εγκλημάτων πολέμου και ως προς την παραδοσιακή δικαιοσύνη χρειάζεται λήψη περισσότερων μέτρων για ισότητα των φύλων, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων η συμπερίληψη των μειονοτήτων στην εθνική ζωή παραμένει ακόμη προβληματική και χωρίς αυτήν δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Η μυσαλλοδοξία Ακόμη υπάρχει κατά των λεσβιών και γενικώ ομοφιλοφίλων. Υπάρχουν επιθέσεις που δεν τιμωρούνται από την αστυνομία. Επίσης, επιθέσεις κατά ε, δημοσιογράφων και γενικώ μαχητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδών επίσης δεν γίνονται και πολύ σεβαστά. Και αυτό αποτελεί πρόσθετο λόγο ανησυχίας. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων συνεχίζουν να είναι χώρες προορισμού δουλεμπορίου, ιδίως για γυναίκες και κορίτσια. Και υπάρχουν πολλοί φραγμοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παιδιά από κοινωνικώς, από κοινωνικώς ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά τσιγκάνων Ρώμα ή ανάπηρα παιδιά υποφέρουν από πολύ περισσότερη άνηση μεταχείριση. Και αυτά είναι λίγα μόνο, όχι όλα από τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω κυρίες και κύριοι ότι θα έπρεπε να αναφέρω ότι όλα αυτά τα θέματα αναλύονται σε περισσότερες λεπτομέρειες όπως και άλλα, μαζί με άλλα, στο χρήσιμο δημοσίευμα έγγραφο που λάβαμε πρόσφατα και που προετοιμάστηκε από το Τμήμα Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης για Εξωτερικά Προγράμματα και ονομάζεται, ονομάζεται λέγω, The Human Rights and Reconciliation in the Western Balkan Countries. Καταλήγοντας κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω κάτι που θα το ξέρετε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η υποεπιτροπή σας πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει θέληση για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά για να είναι αυτή αποτελεσματική χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση και μάλιστα αξιόπιστη πληροφόρηση. Γι' αυτό θα ακούσω πολύ προσεκτικά τι θα μας πείτε σήμερα. Σας καλωσορίζω και εκφράζω και τις ευχαριστίες μου για την απαιτητική εργασία που επιτελείτε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έναν τον ίδιο στόχο να συμβάλλουμε στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να χορηγήσουμε βοήθεια στα θύματα. Είναι δουλειά πολύ δύσκολη και δεν σταματάει ποτέ, αλλά νομίζω ότι όλοι την εκτελούμε με όσο δυνατόν καλύτερη θέληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κούκαν για αυτή την σύντομη αλλά περιεκτικότατη περιγραφή της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή του κόσμου. Ήδη μας είπατε ότι χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τους εμπειρογνώμονές μας και θα ήθελα τώρα πρώτα για 10 λεπτά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νένα Τσέμπεκ του Κέντρου Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και μετά Πέντε λεπτά όλοι οι υπόλοιποι. Και ύστερα η συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη για τους χρόνους αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσει να υπάρξει συζήτηση. Ορίστε πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο ε, από το χρόνο που μου δώσατε. Να σα δώσω ένα δύο παραπάνω στον κανένα. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε να πάρω μέρο σε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Μου ζητήθηκε να σα αναφέρω την κατάσταση πρόοδου τη συμφιλίωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο στοιχείο όσον αφορά το σεβασμό ή μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητήσατε επίση όσο γίνεται περισσότερε πληροφορίε θα σα δώσω όσε μπορώ περισσότερο, αλλά δεν θα είναι όλες καλά νέα. Αν η συμφιλίωση ήταν επιχείρηση, οι επενδυτές θα είχαν φύγει από τα Βαλκάνια εδώ και πολύ καιρό. Εάν ε, ε, θέλουμε να συνεχίσουμε, αν μάλλον η ανθρώπινη φυλή θέλει να συνεχι... θέλουμε να συνεχιστεί, δεν πρέπει να παραγίνει η συμφιλίωση business, αλλά ένα κοπιαστικό, μια κοπιαπιστή προσπάθεια. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και να διασφαλίσουμε ότι ο επωφελούμενοι τη ειρήνη δεν είναι μελλοντικέ γενναίε, αλλά ίσω ακόμα και δικιά μα. Παρακαλώ που να μου συγχωρήσετε που δεν φοράω ροζ γυαλιά για να σα παρουσιάσω μία ρόδινη εικόνα, αλλά θέλουμε σωστέ λύσει, χρειάζονται σωστή διάγνωση. Σωστή διάγνωση σημαίνει να δούμε την πραγματικότητα και όχι τι επιθυμίε μα. Φοβερό πόλεμο, φοβερή πόλεμη γίνανε στα Βαλκάνια, τέσσερι και όλοι με βάση τι αρχέ του 19ου αιώνα που δεν ανήκαν στην Ευρώπη του 20ου αιώνονται στην ε, δημοκρατία. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και ορισμένοι από του κοινικούς μου συναδέλφου, ε, μου το, το περιγράφουν αυτό ως ε, μια ω την εξή σκέψη. Γιατί να είμαι εγώ μειονότητα στη χώρα μου όταν εσύ μπορεί να είσαι μειονότητα στη δική μου. Δηλαδή, σύνορα, επικράτεια, ταυτότητα, θρησκεία ήταν το θέμα. Τι έχουμε σήμερα στην περιοχή, 14 χρόνια μετά από του βασικού πολέμου, 10 χρόνια μετά από το Κωσυφοπίδι και. και, και και ε, ε, από την ε, Φύρωμα. Αυτή τη στιγμή η Σλοβενία είναι η μόνη χώρα που, υπο, που, που μπήκε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία είναι η μόνη που έχει κάποιε πιθανότητε. Αυτέ οι δύο χώρε τσακώνονται για μερικά τετραγωνικά μέτρα γη αλλά και ε, δικαιώματα πρόσβασης στα λιμάνια. Αυτέ οι δύο όμως χώρες θεωρούνται ως λιγότερο επιθυμητός γείτονας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και άλλες χώρες έχουν ζητήσει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τα δημοκρατικά δείγματα που βλέπουμε είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα, πραγματικό, ένα πολύ προσεκτικό μακιγιάζ της πραγματικότητας. Η μετάβαση ε, είναι πολύ σημαντική. Η διαφθορά, το έγκλημα και η έλλειψη ανοχής, η πολιτική ε, ανοχής απέναντι σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς ε, διαφορές είναι προφανής. Η συμφωνία του Ντέιντον θεωρήθηκε ότι θα ήταν μια ασπίδα, αλλά ήταν τελικά ένας πολύ βραχής γάμος ανάμεσα σε τρεις εταίρους, εξ των οποίων οι δύο δεν θέλησαν να ακούσουν ε, δεν, μάλλον δεν αισθάνθηκαν αυτόν τον έρωτα. Πώ μπορεί κανεί να κάνει κάτι με 13 υπουργού παιδεία, για παράδειγμα. 13, διαφορετικά, 13 διαφορετικά υπουργεία πρέπει να επισκεφθώ. Πώ μπορούμε να κάνουμε δουλειά όταν ε, στη χώρα αυτή η, η, εικόνα του γειτονά σου είναι η εικόνα του εχθρού σου. Παρόλε τι προσπάθειε και παρόλα τα εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί για να συγκροτηθεί η Βοσνία, αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μα είναι ένα αποτυχημένο κράτο το οποίο. Ε, ε, αναδίνει μίσος. Αν δεν με πιστεύετε πηγαίνετε στο Μοστάρο που σταμάτησε το 94 οι μάχες. Θα δείτε ότι 15 χρόνια μετά είναι πολύ διαιρεμένοι οι Κροάτες με τους Βοσνίους καθώς και οι λιγοστοί Σέρβοι που επέστρεψαν σε αυτή την πόλη. Είναι ο Δήμος που έχει λάβει περισσότερη βοήθεια κατά κεφαλήν από οποιαδήποτε άλλη κοινότητα στη Βοσνία. Νότιο Δυτικό Μοντενέγρο, το νεό, πιο νεόκοπο κράτος του κόσμου προσπαθεί τώρα να προσδοριστεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία προσβλέπει και τους Ρώσους ολιγάρχες και το κεφάλαιο που το αγοράζουν. Ε, η Σερβία ο νικητής αλλά και, το, και το, ο θήτης και το θύμα των Βαλκανίων. Έχασε το κοσυφοπαίδιο και έχασε και τον δικό της ε, χάρτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι βέβαιη ούτε για τα σύνορά της, ούτε για αυτοτητά της, ούτε για τους στόχους της. Το κοσυφοπαίδιο άλλη νεόκοπη χώρα ε, σύμφωνα με κάποιες από τις χώρες που το αναγνώρισαν. Είναι ένας πολύ, ένα πολύ φτωχό κράτος που πάνω από το 50% είναι η ανεργία και κάθε χρόνο ρίχνει 60.000 ε, νέους άνδρες και γυναίκες χωρίς μια ε, πιθανότητα στο εκατομμύριο να βρουν δουλειά. Δέκα χρόνια μετά από τον βομβαρδισμό τη σερβία από τον ΝΑΤΟ, ακόμα και η μεγαλύτερη αισιοδοξία, ακόμα και οι περισσότεροι αισιόδοξοι έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια τη ανοικοδόμηση ενό πολυεθνικού κοσμοπεδίου. Δεν υπήρχε καταρχήν πολυεθνικό κοσμοπεδίο για να το ανοικοδομήσουμε. Τώρα, για τη Βοσνία, ο Χόντ έβαλε 80.000 τραπεζίτες να υπερασπιστούν τον σταλινισμό του. Ένας, στην Αλβανία, ένας τραπεζίτης δηλαδή κάθε τέσσερις Αλβανοί. είναι μια χώρα που αναγνωρίζεται ως κράτος ως αλλά όχι ως εθνική κοινότητα. Η νότιος ε, σύμμαχός της δεν αναγνωρίζει τώρα το όνομα της ΦΥΡΟΜ και υπάρχει μεγάλη παρακμή όσον αφορά τους, Μακεδο... τους ε, ε, Μακεδόνες και τους Αλβανούς. Ο Χαβιέρ Σολάνα χρειάστηκε να πιάσει τα χέρια των εθνικών ηγετών ώστε να... για να επιτύχει τη συμφωνία της Οχρίδας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μια σκληρή ματιά στην κατάσταση συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Μην με πυροβολήσετε αν δεν σας αλέσετε το μήνυμα. Εγώ είμαι μόνο αγγελιοφόρος. Συ... Ε, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία. Τι περιμέναμε από χώρε που πέρασαν από το φεουδαρχισμό στην απόλυτη μοναρχισμό και από το φασισμό στο κομμουνισμό. Να γίνουν ξαφνικά δημοκρατικές κοινωνίες με ελεύθερο τύπο, ελεύθερες και δίκες εκλογές, ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, να έχουν ένα κρατικό μηχανισμό και, και μη διεφθαρμένη γραφειοκρατία γραφειοκρατία, να, να, να έχουν θεσμικά όργανα που να σημαίνουν κάτι, να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Επιτρέψατε μου να σα θυμίσω Περισσότεροι γνωρίζετε το αστιάκι για του Αμερικανού και του Αμερικα... Εγγλέζου. Έρχεται ο Αμερικανό στον Εγγλέζο και λέει πώ φτιάχνει αυτό το υπέροχο γρασίδι μπροστά στο σπίτι σου και ο Βρετανό λέει χρήχνω του πόρου το ποτίζω και μετά το, ξυρίζω, το κόβω. Και λέει ο Αμερικανό και εγώ το έκανα, αλλά δεν δεν το κατάφερα. Ε, λέει και τότε ο Βρετανό, μα πόσο καιρό το κάνει. Λέει εδώ και τρία χρόνια. Ε, εμεί το κάνουμε εδώ και 300 χρόνια αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και είναι καλύτερο. Αυτή είναι η κατάσταση και εκεί. Υπάρχει κανεί που να πιστεύει ότι πραγματικά μπορούμε να φτιάξουμε τη δημοκρατία πριν να υπάρξει συμφωλίωση μετά από τέτοιου παρακτικού πολέμου. Μια ανόητη φράση που χρησιμοποιούν τα δυτικά ΜΜΕ για τις μετακομμουνιστικές χώρες, ακόμα και για κάποιες μη κομμουνιστικές χώρες όπως η Αϊτή και το Ιράκ, δεν ανικοδομούμε, δεν αποκαθιστούμε τη δημοκρατία εκεί, όπως λένε τα ΜΜΕ. Εμείς προσπαθούμε να φυτέψουμε αυτόν τον ευαίσθητο σπόρο σε πολύ άνεδρο, και καθόλου έφορο περιβάλλον. Ποτέ δεν υπήρξε δημοκρατία στην Αιτή, στην Ρωσία, στην Αλβανία. Οπότε, οπότε ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με άδειο στομάχι δεν μπορούν αυτά να ανθίσουν και η δημοκρατία δεν είναι θέμα του να έχουν μόνο μερικά κόμματα για να διαλέξουν. Άρα και η συμφιλίωση δεν είναι θέμα να υπογράφουμε κάποιε συνθήκε ειρήνη και να λέμε ότι τελείωσε ο πόλεμο. Η συμφιλίωση είναι μια κατάσταση, μια νοοτροπία. Θα παίρνει χρόνο και καθό... πόρο απέχουμε από την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα. Thank you very much, Mr. I think we appreciate... Ευχαριστώ κύριε Σέμπεκ. Ε, ε, εκτιμούμε τα σοφά σας λόγια. Βεβαίως ε, ζήτησα πέντε λεπτά γιατί έχουμε πολλούς εμπειρούς εντός της αιθούσης αλλά δεν θα είμαι τώρα τόσο αυστηρή ε, και ε, εσάς εάν είναι πιο σύντομη η ομιλία σας θα ξεκινήσει πιο γρήγορα η συζήτηση. Η κυρία Κούμιν είναι η Διευθύντρια του Γραφείου για την Ευρώπη το, της ε, Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας στην κατάσταση των ατόμων που ζουν εις, την, τα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως όσον αφορά τους πρόσφυγες και εκτοπισμένους. Θα συνεχίσω την διάγνωση που ανέφερε ο διπλανός μου αναφέροντας ε, το μέγεθος των εκτοπισμών τη δεκαετία του 91. Από το 91 έως το 99 4 ε, εκατομμύρια άτομα ε, εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους πρώτα στην Κροατία και μετά στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και επίσης το Κοσυφοπέδιο. Τώρα, δέκα χρόνια μετά από το τέλος της ε, ε, διαμάχης στο Κοσυφοπέδιο, 17 χρόνια μετά το τέλος του ποέμου στην Κροατία, με τα πρέπει να πω ότι υπάρχουν ακόμη 500.000 άτομα που ζουν εκτοπισμένοι και σαν πρόσφυγες στην περιοχή αυτή. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο μέρος ακόμη των ε, ατόμων που επλήγησαν από αυτούς τους πολέμους. Η διεθνής γνώμη ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για τα, τους πληθυσμούς αυτούς και θα πρέπει να βρούμε λύσεις και αυτό είναι ε, ο πυρήνας για την συμφιλίωση. Ο κύριος Άνιο Κούτρετς πήγε ε, φέτος στην ε, περιοχή, στη Σερβία, στην Κροατία και τους ζήτησε να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη να άρουν τα τελευταία εμπόδια για τους εκτοπισμούς στην περιοχή. Θεώρησε ότι στη Σερβία υπάρχει η πλέον σοβαρή κατάσταση εκτοπισμών, τις οποίες ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει. Ε, και είναι νέος η διοίκηση αυτή αλλά υπάρχουν ακόμη 60.000 πρόσφυγες της ε, Κροατίας που ζουν στη Σερβία υπάρχουν λιγότεροι πρόσφυγες από, την Βοσνία και ένας μικρός αριθμός ε, εκτοπισμένων από το Κωσυφοπέδιο χωρίς να έχουμε τους ακριβείς αριθμούς. Ε, επίσης ενώ δεν το σημειώνουμε το κοστιφοπέδιο ε, έχει μία συνεχή φυγή και αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αιτήσει ετούντων άσυλο από το κοστιφοπέδιο αυξάνονται ενώ είχαν ε, μειωθεί. Τώρα είδαμε ότι μέσα στο εννιάμινο ότι είχαμε περισσότερες αιτήσει από ό,τι πέρυσι όλο το χρόνο. Σχετικά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και ε, το κοσυφοπαίδιο ε, υπάρχουν πολλοί που έχουν εκτοπιστεί και δεν έχουν μπορέσει να επανέλθουν στα σπίτια τους από το 1956 όταν η ε, πρώην Ιουγκοσλαβία ήταν, ε, υποδεχόταν πολλούς πρόσφυγες από το Ανατολικό Μπλοκ ε, και τους προσέραμε ανθρωπιστική βοήθεια τώρα προσπαθούμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο των εκτοπισμών και όπως σας είπα στηριζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στηρίζει το πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής και επαναγκατάσταση αυτών των ατόμων. Ήθελα να σας πω ότι μεταξύ των πιο ευαλώτων τμήματων του πληθυσμού αυτού η ΡΟΜ είναι η πιο ευάλωτοι διότι δεν έχουν καν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σχεδόν παντού και ε, δεν έχουν ε, ουσιαστική τεκμηρίωση διότι οι Ρώμ πολλοί δεν είχαν ποτέ έγγραφα ε, άλλοι έχουν χάσει τα έγγραφα άλλοι δεν έχουν καταγράψει τη γέννηση των παιδιών τους ή στο παρελθόν ή δεν το κάνουν καν ακόμη και ε, πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέψει στους δρόμους να αποκτήσουν ε, ε, τα έγγραφα που χρειάζονται και να καταγραφούν γιατί αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να επιληθεί το πρόβλημά τους. Όπως ε, είπατε δεν έχουμε χρόνο κυρία Πρόεδρε, αλλά ίσως καλό θα ήταν να τονίσω εδώ τρία πράγματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε κατά προτεραιότητα. Πρώτα ε, μία λύση για τους Κροάτες πρόσφυγες που ζουν στη Σερβία και χρειαζόμαστε εκεί την ε, συμμετοχή των αρχών για να αποκτήσουμε ακριβείς στατιστικές για τους ποιους παραμένουν στη Σερβία ή έχουν επιστρέψει επιστρέψει στην Κροατία. Όποιος θελήσει να επιστρέψει στην Κροατία πρέπει να βοηθηθεί να το πράξει. Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες και πολλά εξατώνται από το δικαίωμα παραμονής που έχουν οι ε, Κροάτες ή είχαν την εποχή της σοσιαλιστικής δημοκρατίας και ζητούμε από την κυβέρνηση της Κροατίας να αποζημιώσει τα άτομα αυτά και να τους βοηθήσει να επανεγκατασταθούν. Ε, ορισμένοι θέλουν όμως να παραμείνουν μονίμως στη Σερβία, πολλοί το έχουν πράξει ήδη και θα έπρεπε να βοηθηθούν στο θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν εκεί αν το επιθυμούν. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα των ε, ε, προσφύγων του κοστιφοπεδίου που ζουν ε, εις τις διάφορες άλλες δημοκρατίες. Το, το ερώτημα είναι αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν. Πότε θα αισθανθούν ασφαλείς να επιστρέψουν και αν όχι μπορούμε να, βοηθήσουμε, να τους βοηθήσουμε να ενσωματωθούν στην περιοχή όπου μένουν και να βοηθηθούν για να μπορέσουν να εγκατασταθούν. Τέλος πρέπει να βρούμε λύσεις ε, για τους Σέρβους και Ρόμ που έχουν ε, ε, μετατοπιστεί στο Κωσυφοπαίδιο ως επτοπλίστων πρόκειται για Αλβανούς οι οποίοι επιστρέφουν γρήγορα αλλά οι μειονότητες έχουν, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και είναι ένα πρόβλημα που έχουμε και στην Ευρώπη διότι οι περισσότεροι εκ των οποίων απορρίπτεται γίνεται η αίτηση ασύλου παραμένουν πολύ προβληματικοί. Έχοντας λοιπόν επί δύο δεκαετίες διαπιστώσει τις εκτοπίσεις στα Δυτικά Βαλτάνια πρέπει να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να ζητήσουμε από όλου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα γειτονικά κράτη, από την κοινωνία των πολιτών να βοηθήσουν να επιληθεί αυτή η δεκαετία ε, των εκτοπισμών. Ευχαριστώ. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σας έχει βοηθήσει και τώρα θα απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον υπεύθυνο ε, ε, για θέματα... Αλβανίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ευγνωμοσύνη μας για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, γιατί χρειαζόμαστε την ε, βοήθεια της Επιτροπής σας για να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Επίσης, το έγγραφο που προετοίμασε η Γραμματεία νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων είναι θέματα που συμπεριλαμβάνονται στους ενταξιακούς στόχους της Κοπεχάγης ενώ τα θέματα των προσφύγων είναι τμήμα της διαδικασίας σταθεροποίησης. Γι' αυτό στην Κομισιόν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα αυτά και παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως την τελευταία μας έκθεση τον Οκτώβριο. Επίσης χορηγούμε χρηματική βοήθεια είναι προφανές. Φυσικά συνεργαζόμαστε με την υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και άλλες οργανώσεις. Λοιπόν, τι αξιολόγηση κάνουμε γενικά. Παρά τις κοινέ μας προσπάθειες, δηλαδή με την υπάτη αρμοστία, το επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ακόμη ανησυχητικό. Όχι τόσο διότι λόγω του νομικού πλαισίου διότι το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο ε, δημιουργείται σιγά σιγά στις περισσότερες χώρες. Σε μερικές μάλιστα σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Έχουν εγκριθεί προγράμματα και στρατηγικές για την προστασία των μειονοτήτων, νομοθεσία για ίση μεταχείριση, έχει εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθεί ως τμήμα των συνεννοήσεων για τις θεωρήσεις. Και αυτά είναι όλα πολύ θετικά. Αλλά το θέμα είναι μάλλον η διαφορά μεταξύ των νομοσχεδίων και της εφαρμογής τους, του νόμου και της επιβολής, η εφαρμογής του νόμου. Μερικές φορές δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Άλλες φορές λείπουν τα χρήματα. Και φυσικά η οικονομική κρίση και οι περικοπές στον προϋπολογισμό, στους προϋπολογισμούς προσθέτουν δυσκολίες. Για να είμαι σύντομος λοιπόν γενικότερα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν μιλήσουμε για τους πρόσφυγες και την συμφιλίωση θα έλεγα ότι το κυριότερο θέμα που μας ανησυχεί είναι η κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Πολύ συχνά γίνονται θύματα βίας Άλλο θέμα είναι οι αντιομοφιλόφιλες τάσεις, οι ομοφοβικές τάσεις και οι απειλές ή βιοπραγίες κατά μαχητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως δημοσιογράφων. Αυτό φυσικά περιορίζει το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η μήκη όμικρον. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το δουλεμπόριο, το εμπόριο λευκής σαρκός, και μία μειονότητα που υποφέρει περισσότερο από τις άλλες είναι η Τσιγκάνη, η Ρώμα. Φυσικά αυτό είναι, αυτά όλα είναι πολύ χειρότερα για πρόσφυγες, ιδιαίτερα για γυρεότερους που εδώ και 15 χρόνια ζουν σε πολύ άσκημες συνθήκες. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδο στην Κροατία, στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, αλλά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δεν συμβαδίζουν καθόλου με τις ανάγκες που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες. Τώρα, αναχώρα. Στην Κροατία νομίζουμε ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι όσοι πρόσφυγες θέλουν να επιστρέψουν στην Κροατία έχουν κάποιο πρόγραμμα υποδοχής αλλά σε πολλές χιλιάδες περιπτώσεων, όπως είπε και η κυρία Κούμιν, τα πράγματα δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Στο λεγόμενο κεφάλαιο 23 των ενταξιακών συνεννοήσεων, που δεν έχει ακόμη ανοίξει, πρόκειται όμως να ανοίξει, έχουμε βάλει μεταξύ των κριτηρίων και την αμοιβαία αναγνώριση των συνταξιοδοτήσεων και άλλα συγκεκριμένα θέματα για τους πρόσφυγες και ελπίζουμε οι όροι αυτοί που έχουμε θέσει να είναι αποδοτικοί και να καταλήξουν σε, σε κάτι το θετικό. Στην ε, Πουγουδουμού το θέμα, το πρόβλημα είναι πιο περιορισμένο, όχι μόνο γιατί είναι λιγότεροι οι πρόσφυγες, αλλά επίσης και λόγω της προόδου που έχει γίνει για την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπάρχουν ακόμη λήψεις και χάσματα μεταξύ των νόμων και της εφαρμογής του. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη έχουμε χορηγήσει βοήθεια για στέγαση και το σημαντικότερο είναι ότι έχει ε, γίνει η επεξεργασία μια στρατηγικής στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με τη βοήθεια τη Υπάτη Αρμοστία, όπου 250 εκατομμύρια έχουν χορηγηθεί, θα χορηγηθούν 250 εκατομμύρια ευρώ για την επιστροφή προσφύγων. Αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί το πρόγραμμα γιατί, γιατί υπάρχει διαφωνία ως προς το κατά πόσο θα πρέπει τα χρήματα αυτά να δοθούν αποκλειστικά για επιστροφέ ή και για την η υποδοχή ή υποβοήθηση προσφύγων που δεν θέλουν να επιστρέψουν. Δεν έχει ακόμα υπάρξει συμφωνία λοιπόν και το πρόγραμμα αυτό, η στρατηγική αυτή είναι ακόμη παγωμένη στο, στη Βουλή. Μετά από αυτά που είπε ο κ. Σεμπέκ για το Μουστάρ, ε, θέλω να προσθέσω το εξής. Πώς μπορεί κανείς να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση όταν όχι μόνο στο Μοστάρ αλλά και αλλού υπάρχουν δύο σχολεία στο ίδιο κτίριο δηλαδή. Παιδιά μουσουλμάνων ή καθολικών δεν παίζουν ποτέ μαζί ούτε πηγαίνουν στην ίδια τάξη. Πώς μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση λοιπόν. Στο Μαυροβούνιο το κύριο θέμα είναι οι εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγες ιδίως από το Κωσυφοπαίδιο το θετικό είναι ότι στα πλαίσια του διαλόγου για τις θεωρήσεις το Μαυροβούνιο τώρα κάνει μια νέα απογραφή των εκτοπισμένων για να τους δώσει, να τους χορηγήσει ένα επίσημο καθεστώς και να μπορέσουν έτσι να ζητήσουν ε, να κάνουν αιτήσει για στεγαστική βοήθεια και άλλα, άλλα είδη. Οι σχέσεις Κωσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου θα βοηθήσουν με τα πράγματα για τους εκτοπισμένους. Για τη Σερβία δυστυχώς δεν έχουμε πολλά αξιόπιστα στοιχεία για τους πρόσφυγες ή εκτοπισμένους, αλλά ξέρουμε ότι τουλάχιστον 5.000 ακόμη ζουν σε συλλογικά κέντρα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα οι τσιγκάνοι και πολύ λίγοι έχουν επιστρέψει στο κοσυφοπαίδιο. Νομίζω ότι οι αριθμοί για το 2008-2009 είναι περίπου 900 μόνο. Γιατί όχι περισσότεροι, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης, ούτε στέγασης. Εμείς διευκολύνουμε τις επιστροφές, χρηματοδοτούμε στεγαστικά προγράμματα αλλά δεν επιστρέφουν. Δεν θέλουν να επιστρέψουν δηλαδή. Και στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα ετοιμάζονται προγράμματα για επιστροφές, χωρίς να υπάρχει διάλογος βέβαια, και δεν ξέρουμε αν τα δύο προγράμματα θα ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο, αλλά ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διάλογο ώστε τα δύο αυτά προγράμματα της Πρίστινας και του Βελιγραδίου να συνδυαστούν. Λοιπόν, η επιστροφή και επανεγκατάσταση προσφύγων και εκτοπισμένων έχει καθυστερήσει, έχει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες και η διαδικασία του Σαράγεβου που υπετίθετο ότι θα έβρισκε κάποια λύση για αυτούς έχει σχεδόν σταματήσει. Γι' αυτό δεχόμαστε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Βελιγραδίου να οργανωθεί μια υπουργική διάσκεψη και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε στη διοργάνωσή της. Η διαδικασία σταθεροποίησης είναι απαραίτητος παράγοντας βέβαια για τη συμφιλίωση. Πώς μπορεί να υπάρξουν καλές σχέσεις μεταξύ χωρών αν χιλιάδες άνθρωποι ζουν ακόμη υπό συνθήκες προσφυγιάς και εκτοπισμού. Και με τι ελεύθερη, τι ελεύθερη επιλογή, με ελεύθερη επιλογή να επιστρέψουν βέβαια θέλουμε, όχι υποχρεωτικά. Να μπορούν να μείνουν αν θέλουν στη χώρα όπου διάλεξαν να πάνε. Και κατ' εμάς υπάρχει και μια, ένας άλλος όρος για τη συμφιλίωση, να δικαστούν οι εγκληματίες πολέμου. Όπως ξέρετε αυτό είναι ευθύνη του ποινικού δικαστηρίου και των εθνικών, του διεθνούς ποινικού και των εθνικών και εμείς έχουμε ζητήσει τρεις Έχουμε θελήσει να εφαρμόσουμε τρεις τρόπους συνεργασίας. Χρηματικά, για εκπαίδευση δικηγόρων κλπ. Δεύτερον, μέσω της χορήγησης χρηματικής βοήθειας σε εθνικά δικαστήρια στην Κροατία, στη Βοσνία, Ζεγοβίνη, στη Σερβία και νομίζω ότι υπήρξε κάποια πρόοδος ιδιαίτερα όμως στο Σεράγεβο υπάρχουν ακόμη χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις Επίσης πολύ δύσκολο θέμα για τους εθνικούς εισαγγελείς και δικαστές είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χωρών για τις εκδόσεις. Δεν υπάρχει συμφωνία αμοιβαίων εκδόσεων. Πολλές περιπτώσεις δεν ανοίγουν καν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει έκδοση των εγκληματιών και πολέμου και κοινών ποινικών. Επίσης στηρίζουμε τρίτον πάλι χρηματικά τις τοπικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που αναλαμβάνουν να βρουν και να πούν την αλήθεια. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι τελείως απαραίτητο για τη συμφιλίωση και για την λεγόμενη μεταβατική δικαιοσύνη. Υποστηρίζουμε λοιπόν και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στο Σεράγεβο και στο Βελιγράδι που όπως είπα, ψάχνουν να βρουν την ιστορική αλήθεια. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση. Έτσι πιστεύω. Και αυτό είναι το μάθημα που πήραμε από την ιστορία και της ευρωπαϊκής κοινότητας. Οι μήκοι όμικρον σε όλες αυτές τις χώρες έχουν αναλάβει μια καινούργια πρωτοβουλία που λέγεται Ρίκομ θέλουν να πιέσουν τις κυβερνήσεις <coughs> να είναι λίγο πιο πρόθυμες για τις διώξεις των εγκληματιών και για τη συμφιλίωση ώστε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη και να μπορέσουν οι μελλοντικές γενιές να μάθουν, να πάρουν μαθήματα από το παρελθόν. Και αυτό το υποστηρίζουμε. Και στις αρχές Δεκεμβρίου οργανών, συνοργανών, συνδιοργανώνουμε σεμινάριο εδώ στις Βρυξέλλες με αυτές τις οργανώσεις. Νομίζω εδώ δεν υπάρχει καθόλου χώρος και χρόνος για εφησυχασμό. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν θα συνεχίσει να το πράττει και υπολογίζει και στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των οργανώσεων που είναι παρούσες εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε πως ε, η διαδικασία είναι σε πολύ καλά χέρια στην Επιτροπή και μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα της μεταβατικής δικαιοσύνης ο επόμενο ομιλητή είναι ο κ. Μπογκδάν Ιβανίσεβιτ, που αντιπροσωπεύει το Διεθνέ Κέντρο για τη μεταβατική μετάβαση μάλλον στη δικαιοσύνη στο Βελιγράδι. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο οργανισμός μας, το Διεθνές Κέντρο για την ε, Μεταβατική Δικαιοσύνη, έχει ως έδρα του τη Νέα Υόρκη. Εγώ ζω στο Βελιγράδι για τους σκοπούς της αποστολής. Δεν έχω επιλογή από το να είμαι πολύ σύντομος ε, λόγω των χρονικών σας περιορισμών, αλλά θα είμαι ακόμη συντομότερος δεδομένου ότι ο κύριος Μιρέλ ιδιαίτερα στο δεύτερο ήμιση της παρουσίασής του, ανέφερε διάφορα πράγματα τα οποία θα έλεγα και εγώ. Και με θάρρυνε που άκουσα από εκείνον τα σχετικά, διότι πραγματικά είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Και αν έχω χρόνο θα σας πω και εγώ δύο λεπτομέρειες. Όταν μιλάμε για την μεταβατική δικαιοσύνη, συνήθως μιλάμε για τέσσερις στάνταρ μηχανισμούς, που είναι οι ποινικέ διώξεις, οι επανορθώσεις, οι, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις και η αναζήτηση της αλήθειας, όπου ανήκει και αυτή η πρωτοβουλία Ρέκομ. Στην παρουσίασή μου θα μιλήσω για αυτούς τους τέσσερις πυλώνες χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για το πώς κάθε χώρα τα πάει για κάθε λεπτομέρεια. Εν γέννη, 15, εδώ και 15 χρόνια το θέμα της μετρατικής δικαιοσύνης έχει μονοποληθεί από το θέμα της ε, δίωξης ε, για εγκλήματα πολέμου, κυρίως για την πρώην Ιουκοσλαβία, αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει θέσει αυτούς τους όρους. Το Διεθνές ε, Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία στην Χάγη έχει διώξει πολιτικούς ηγέτες προτίμαζοντας το έδαφος για εθνικές δίκες για εγκλήματα πολέμου όμως δεν ε, μπόρεσε και δεν μπορούσαμε και να αναμένουμε να συμφιλιώσει τα ε, διάφορες εθνοτικές ομάδες, πράγμα που μας ε, ανέφερε και ο κύριος Σάντεκ με ιδιαίτερη φράδια. Όσον αφορά τις προσπάθειες ε, για την ε, δίωξη των ε, κλιμάτιων πολέμου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ξεκίνησαν στην αρχή αυτής της δεκαετίας με την αναχώρηση από την αρχηγία των ηγετών της διάρκειας του πολέμου στην Κροατία και τη Σερβία. Ένδειξη για την πρόοδο που έχει σημειωθεί είναι ότι ο αριθμός των δικών που, γίνεται, ε, που γίνονται κατά της, ε, των ηγετών είναι την πλειοψηφία από καθοδηγούνται από τον ίδιο τον πληθυσμό. Όμως παρά την πρόοδο, μόνο ένα μικρό ποσοστό των εγκληματιών πολέμων έχουν δικαστεί ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Υποστήριξη από τις πολιτικές δομές για την δίωξη μελών της ε, πλειοψηφικής, ε, του μεγαλύτερου μάλλον πληθυσμού σε κάθε χώρα είναι περιορισμένη. Μια σημαντική θετική εξαίρεση στη Βοσνία είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη, πράγμα το οποίο μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι το ειδικό τμήμα για τα εγκλήματα πολέμου στο Σαράγεβο, στο εισαγγελικό γραφείο, είναι ένα υψηλό επίπεδο θεσμικό όργανο όπου οι διεθνεί αρχέ συνεργάζονται με τι βοσνιακέ και στα 3,5 χρόνια εντατική λειτουργία. λειτουργία δηλαδή της, του ειδικού αυτού τμήματος στον Άρη Πάγο της Βοσνίας Ερζογοβίνης έχουν, εκδικαστεί 30 τελεσίδικες ε, δίκες, ε, έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις και προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι ένα ρεκόρ για όλες τις χώρες ε, εδώ και 15 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου της Βοσνίας και της Κροατίας. 200 υποθέσεις έχουν τελικά εκδικαστεί σε όλες τις χώρες. Είναι μια προς, κατά προσέγγιση αριθμός είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Βεβαίω, ε, ο ρυθμό στον οποίο εκδικάζονται όλε αυτέ οι υποθέσει είναι ιδιαίτερα, είναι, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό λόγω των χιλιάδων εγκλημάτων πολέμων που έχουν διαπραχθεί ναι. κατά τη διάρκεια των ε, του πολέμου στην περιοχή. Τώρα, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι μόνες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε μεταγιουγκοσλαβική χώρα με στόχο την ε, απομάκρυνση των παραβιαστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν αυτές που ε, ε, έγιναν το 1999 με 2002 στη Βοσνία για την αστυνομία και 2002 και 2004 για το δικαστικό σώμα δικαστική μεταρρύθμιση. Τώρα, η δικαστική μεταρρύθμιση εν γέννη έγινε αντιληπτή ω ε, σχετικά ικανοποιητική και επιτυχής γιατί μείωσε τον αριθμό των ε, ανθρώπων που βρίσκονταν σε υψηλέ θέσει, χωρί να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Στη Σερβία ένα νόμο για την ευθύνη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υιοθετήθηκε το 2003, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. η προετοιμασία στην πρώην Οικοσλαβία, τόσο οι υλικέ όσο και οι συμβολικέ προετοιμασίε, έχουν γίνει βασικά από τα μέλη των ε, μεγαλύτερων εθνικών, εθνοτικών ομάδων, ενώ η διαδικασία είναι ακόμα στην αρχή όσον αφορά τι μειονότητε, ε, δηλαδή του εχθρού, του ε, αντιπάλου του πολέμου. η αρχή της αλληλεγγύης για τα θύματα και η αρχή της κατάχρησης σχεδόν της επανόρθωσης μάλλον για κατάχρηση είναι σχεδόν απούσα από όλη τη διαδικασία. απώλεια ζωής ή ε, ζημιά, βλάβη στην υγεία του ανθρώπου, αυτά πολύ σπάνια έχουν αποζημιωθεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ε, εθνοτική βία μπορεί να έχει ασχηθεί ε, κυρίως από, το στρατιωτικό, τους και έτσι δίνεται περισσότερη προτεραιότητα σε αυτούς. Δεν υπήρξε πραγματική σύσταση επιτροπή για την αναζήτηση τη αλήθεια σε οποιαδήποτε από τι χώρε τη επικράτεια τη πρώην Ιουγκοσλαβία. Η μόνη που τουλάχιστον επισήμω θεσπίστηκε και υπήρξε είναι η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης στην τότε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας που θεσπίστηκε το 2001 αλλά διαλύθηκε μετά από ένα χρόνο χωρίς να πετύχει τίποτα. Τη απουσία σύσταση τέτοιων επιτροπών, το ICTY και σε κάποιο βαθμό και τα τοπικά δικαστήρια, καθώς και κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ΜΜΕ αλλά και ιστορικοί, συνέβαλαν στην αποκατάσταση της αλήθειας στην περιοχή και ως προς αυτό οι προσπάθειες δύο ΜΚΟ θα πρέπει να τονιστούν. Είναι το ερευνητικό κέντρο στη Σαράγεβο, και το αντίστοιχο του Βελιγραδίου και τα δύο έκαναν ε, μητρώα ανθρωπίνων απολειών με τα ονόματα όλων των θυμάτων. Η πραγματική πρόκληση στην πρώην Ιγκοσλαβία είναι να βρεθεί ένας τρόπος για να θεσπιστούν τα γεγονότα, ε, ε, αλλά με τρόπο που να γίνει αποδεκτός από το κοινό τα εγκλήματα πολέμου και άλλες προσπάθειες για να καταγραφεί αλήθεια για το παρελθόν δεν αναγνωρίστηκαν και δεν επέφεραν πρόοδο στην ε, ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες εθνωτικές ομάδες στην περιοχή. Και γι' αυτό, σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε αυτή η ιδέα για την ε, Επιτροπή ε, αλήθειας, ανέβρεσης μάλλον, αναζήτησης της αλήθειας από τις διάφορες ΜΚΟ. Αυτή τη στιγμή ένας μη κυβερνητικό συνασπισμός 230 ε, περίπου οργανώσεων καθημερινά κάνει συναντήσεις που αποτελούν τμήμα της διαδικασίας διαβούλευσης, στόχος της οποίας είναι να θεσπιστεί αν υπάρχει ζήτηση στην κοινωνία από την κοινωνία των χωρών να αναθεσπιστεί μια επίσημη Επιτροπή Αναζήτησης της ε, Αλήθειας. Ε, η ιδέα είναι να υποβληθεί στις κυβερνήσεις των περιοχής μέχρι το τέλο του 2010 ε, μια επίσημη, ένα επίσημο αίτημα το οποίο θα στηριχθεί από υπογραφές διαφόρων ανθρώπων από την περιοχή ώστε να δημιουργηθεί από κοινού μια τέτοια επιτροπή. Γνωρίζω πως δεν έχω χρόνο να επιμείνω σε αυτό. Πάντως είναι μια διαδικασία η οποία αξίζει να υποστηριχθεί. Yes. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίες όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και είναι σωστό που τις συζητάμε σήμερα που γιορτάζουμε την πτώση του τείχους του Μπερολίνου γιατί έτσι στο Βερολίνο είδαμε να πέφτουν δύο δικτατορίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα θα γίνουν οι δηλώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Είναι δύο οι εκπρόσωποι, θα μοιράσουν το χρόνο τους, δύσκολο πράγμα το ξέρω, αλλά ελπίζω να μας αφήσετε χρόνο και για τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω εγώ, η Σάιαν Jones. Θα πω τα μισά να πει τα άλλα μισά ο συνάδελφός μου. Λοιπόν, θα περιοριστώ σε τρεις πτυχές του θέματος. Ελπίζουμε οι διεθνείς αμνηστία να καταφέρει να επηρεάσει τα πράγματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει εφαρμογή τους και όχι απλώς καθορισμό στα χαρτιά. Η διεθνής αμνηστία αυτό ζητάει να πετύχει. Έτσι ώστε να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων που έχουν υποφέρει από παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Το πρώτο θέμα που θα θίξω λοιπόν είναι οι εξαφανίσεις και απαγωγές. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε ότι το γεγονός ότι οι αρχές δεν καταφέρνουν να κάνουν τις έρευνες για τους εξαφανισθέντες είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σχετίζεται με τα σημεία που αφορούν τα βασανιστήρια στη Σερβία, στην Κροατία, στη Βοσνία, στο Βοσιφοπέδιο και στο Μαυροβούνιο έχουμε τουλάχιστον 50 με 60 χιλιάδες ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα αγαπημένα των πρόσωπα. Έχουμε εδώ ένα φυλάδιο που λέγεται το βάρος του παρελθόντος και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια αυτό είναι το πρόβλημα πρέπει να έχουν το δικαίωμα όλοι να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι συγγενείς τους. Το μόνο, η μόνη περίπτωση που διαπιστώσαμε να γίνεται κάτι για τους εξαφανιστέντες ήταν στο Μαυροβούνιο πέρυσι όπου είχαν προβλεφθεί αποζημιώσεις για ορισμένους που είχαν εκδοθεί στις αρχές της Ρεπούμπλικας Σέρψκας. Υπάρχει μια σειρά συστάσεων που θα αφορούσαν ιδιαίτερα τη χώρα αυτή αλλά θα μπορούσαν να ισχύουν και για όλες τις υπόλοιπες χώρες όπως η υποστήριξη που μπορεί να δοθεί στο Δικαστήριο ε, Εγκλημάτων Πολέμου για τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο, αλλά θα θέλαμε επίσης να υπάρξει και συνέχιση της στήριξης της αποστολής αυτής, διότι υπήρξε κάποια πρόοδος στην δίωξη των όσων έχουν οδηγήσει τον κόσμο να αλλάξει χώρα. Να συνεχίσουμε λοιπόν τη στήριξη των προσπαθειών αυτών ώστε σε ολόκληρη την περιοχή αυτή να δοθούν τουλάχιστον αποζημιώσεις για τους εξαφανισθέντας ή τους αγνοούμενους. Όσοι στα Δυτικά Βαλκάνια ζητούν την ε, εκδίκαση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου διώκονται τελικά. Στη Σερβία τρεις γυναίκες μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων η Νατάσα Κάντιτς, Σόνια Μπιζέρκα και η Μπίλιανα, δεν λέει το επίθετο η ομιλήτρια, είναι γνωστές περιπτώσεις σε όλους σας μάλλον. Έχουν κατηγορηθεί ότι υποστηρίζουν την ένταξη στην Ένωση. Έχουν κατηγορηθεί ότι ζητούν ευθύνες, να αποδοθούν ευθύνες για τους εγκληματίες πολέμου. Πριν από μερικά χρόνια υπήρξε το έγγραφο κατευθυντήριες γραμμές για υποψήφιες χώρες και στη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο, την Κροατία, τη Βοσνία ζητήθηκε να εφαρμόσουν τις κατευθυντήρες αυτές γραμμές για να διασφαλιστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε όταν κανείς απειλείται από διώξεις τέτοιου είδους ή όταν απαγορεύεται η Gay Pride στο Βιλιγράδι σε τέτοιες περιπτώσεις όλες οι πρεσβείες των χωρών μελών να διαμαρτύρονται ομόφωνα για να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος. Χαίρομαι που οι εκπρόσωποι εδώ και της Κομισιόν και της ΥΠΑ της Αρμοστίας τόνισαν ότι αυξάνονται συνεχώς οι αριθμοί των προσφύγων. Εμείς θα θέλαμε να ξεπεράσουμε λίγο τις προτάσεις τους και να ζητήσουμε από τις χώρες της Ένωσης που θέλουν να συνάψουν διμερείς συμφωνίες με το κοσυφοπέδιο ας πούμε να μην δέχονται τις επιστροφές τσιγκάνων, δεν νομίζω ότι οι Σέρβοι έχουν ζητήσει να επιστρέψουν, με το ζόρι. Αλλά οι επιστροφές να γίνονται και θελοντικά αλλά και με τη διάθεση των απαραίτητων υλικών μέσων. Η Κροατία είχε πει αν έχει αρκετά χρήματα μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υποδοχής ίσως και στο Μαυροβούνιο να κατορθωθεί να επιστραφούν πρόσφυγες στο Κωσυφοπαίδιο γιατί αλλά οι περισσότεροι τσιγκάνοι πρόσφυγες από το Κωσυφοπαίδιο ζουν σε χώρες της Ένωσης Θα έπρεπε οι αρχές του κοσυφοπεδίου να βοηθηθούν να δημιουργήσουν τις υποδομές που να επιτρέψουν τις επιστροφές. Αλλιώς θα παραμείνουν σε άλλες χώρες όπως τη Σερβία. Ανά μερικά συγκεκριμένα πράγματα που συστήνουμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. για να υπάρξουν αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Jones. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, άπαξ και μιλήσατε για τις κατευθυντήριες γραμμές της προασπίσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι δεν ξέρουν πώς οι αντιπροσωπείες εφαρμόζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές χωρίς σχόλιο ή απο... χωρίς ε, μικρόφωνο η απάντηση δυστυχώς. Πολύ ωραία γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία για την καλή διακυβέρνηση και για τις εξωτερικές μας αποστολές. Το έχω συζητήσει και μου ελέγχθη ότι υπήρξαν ορισμένα παράπονα για ορισμένες από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και ε, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνει ορισμένες ε, εξετάσεις ε, για να το έχετε υπόψη σας θα πρέπει να έχουμε χρόνο και για όσους από τους παρισταμένους ε, ζήτησαν να ε, παρέμβουν η κυρία Ντεκάιζερ πρώτα και ε, άλλοι όσους προλάβουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω και τον άλλο συνάδελφο, φίλο τουλάχιστον από την Διεθνή Αμνηστία. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσει να παρέμβει αργότερα. Βεβαίως όταν ακούμε τους διάφορους συνομιλητές μας ε, διαπιστώνουμε ένα παράδοξο διότι όντως η κατάσταση στην οποία περιγράφουν είναι και περίπλοκη και σχετικά δυσάρεστη από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία να την οικοδομήσουμε διότι ποτέ δεν έχει υπάρξει σε αυτές τις χώρες. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρετε ότι Πολλοί Ευρωπαίοι έχουν χάσει την όρεξή τους για τη διεύρυνση, λένε πρέπει να σταματήσουμε τις διευρύνσεις. Αυτό ακούω τουλάχιστον στο δρόμο. Και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και τα Βαλκάνια αποτελούν έναν γεωγραφικό χώρο όπου ε, ρητός ή εμέσως πιστεύουμε ότι έχουμε μία υποχρέωση να επεκταθούν προς τα Βαλκάνια. Αλλά αν χρειαζόμαστε 600 ή 800 χρόνια για τον καζόν και για τη δημοκρατία δεν μπορούμε να δεχθούμε στην Ευρώπη χώρες όπου η δημοκρατία δεν είναι κάπως σταθεροποιημένη. Είναι πολύ δυσάρεστο. Πώς μπορούμε λοιπόν να ε, διερευνήσουμε θέματα που λειτουργούν σωστά και πολύ καλά ο κύριος Μιδιέλ ανέφερε ό,τι έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ έχω μία σύντομη ερώτηση. Για μένα το κοσυφοπαίδιο είναι μία σχολική περίπτωση. Είναι ε, κάτι που έχει καταρτιστεί χωρίς να αναγνωριστεί από την Ευρώπη ε, ένας μικρός χώρος ε, τον οποίον, από τον οποίο περιμένουμε πολλά διότι δημιουργείται τεχνητά. Και μετά είπαμε Έχουμε ήδη προβλέψει εκεί ε, δαπάνες, χρηματοδοτήσεις και ε, όταν ε, είδα ε, ποιοι φάκελοι ε, πρόκειτο να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη μεταξύ εγκληματιών και εγκληματιών πολέμου θα ήθελα κάποιος να μπορέσει να μου πει τελικά τι έγινε ποια ήταν η συμφωνία η οποία επετεύχθη και ποιο ήταν το επιπρόσθετο κρέος, κέρδος που μας κόστησε πολλά και που επιτύχαμε στο Κωσυφοπέδιο διαφορετικά πρέπει να απογοητευτούμε πλήρως. Τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω, τι άτομα, τι ε, πόρους πρέπει να διαθέσουμε επιπλέον. Ε, θα ήθελα να μου πείτε αν λειτουργεί, αν έχει λειτουργήσει, εάν πρόκειται να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ κυρία Ντεκάιζερ. Ο κύριος Πρόντινο, επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε ήθελα να ευχαριστήσω Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέμπεκ ιδιαίτερος και τον κύριο Ιβανή Σεβίτσο ε, για τις παρεμβάσεις τους που ήταν πραγματικά πολύ ρεαλιστικές. Και εγώ διερωτώ με αν μπορεί να γίνει για ολόκληρη την πρώην Ιουγκοσλαβία μια διαδικασία αλήθειας και συμφιλίωσης. Γιατί πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να γίνει. Όλος ο κατακαιρματισμός της πρώην Ιουγκοσλαβίας πραγματικά εμποδίζει την εξέβρεση της αλήθειας. Γιατί το πλαίσιο της πρώην Ιουγκοσλαβίας παραμένει κατακαιρματισμένο. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και στη δικασία διεύρυνσης θα πρέπει να, να συστήσουμε εκ νέου το πλαίσιο της πρώην Ιουγκοσλαβίας όσο γίνεται περισσότερο. Κατά κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε όχι μόνο τα κατάλληλα όργανα, δομές, νόμους κτλ. σύμφωνα με τις δικές μας προδιαγραφές, αλλά διαδικασία διεύρυνσης να μπορέσει να επινοήσει μια διαδικασία ε, και συμφιλίωσης. Γιατί τα δύο πράγματα θα πρέπει να προχωρήσουν μαζί και πιστεύω πως θα πρέπει να αναζητήσουμε κάθε τρόπο για να, να συστήσουμε την ενιαίο χαρακτήρα του σκηνικού της βίας διότι Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πραγματική διαδικασία ειρήνευσης και πραγματική συμφιλίωσης. Και νομίζω πως και η δραστηριότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου, του, προ... ποινικού Διεθνούς Δικαστηρίου για την πρώην Ιγκοσλαβία, προχώρησε στο να θεσπίσει προσωπικές ευθύνες, που είναι απαραίτητο, αλλά σκίασε έτσι τη διαδικασία αλήθειας και συμφιλίωσης που είναι η διαδικασία την οποία χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση. Διαρωτώ με λοιπόν μήπως είναι δυνατόν να ε, γίνει ή και να συνδεθεί η διεύρυνση με την ανασύσταση του πλαισίου της πρώην Ιουκοσλαβίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο πραγματικά αλήθειας για να γίνει και η συμφιλίωση. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ακόμα μιλητές. Τον Αντιπρόεδρο Ζέμκε και μετά την κυρία Γιαννάκου. Κύριε Ζέμκε. E, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις πληροφορίες, διότι ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία και θα έλεγα μάλιστα ότι πρόκειται και για μια σαφέστατη περιγραφή της κατάστασης. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για τη συζήτηση, όλο και λιγότερο χρόνο έχουμε. Το ρολόι προχωράει γρήγορα, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω την προσοχή σε ένα ερώτημα και αυτό σχετίζεται με το όσο είπε η κυρία Ντεκάιζερ και ο κύριος Πρόντι. Ως ευρωβουλευτές έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δίλημα, να κάνουμε μια επιλογή κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή όχι της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίζει να ευδιευρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η οχι της διευρυνσης της ευρωπαικης ενωσης θελουμε να συνεχιζει να ευδιβρυνεται η ευρωπαικη ενωση αλλα αυτη η συζητηση μας δείχνει πως κυρίως όταν πρόκειται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε κυρίως για δύο κράτη, την Ισλανδία όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και την Κροατία που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας όσον αφορά τη διεύρυνση της Ένωσης. Και γι' αυτό και έχω αυτή την απλή ερώτηση. Τι πιστεύετε για την κατάσταση της κρατίας, Πώς την αξιολογείτε αυτή την κατάσταση. Γιατί με βάση τις πληροφορίες που ακούσαμε σήμερα, Μα λέτε πως δεν υπάρχει χώρος για τους πρόσφυγες, πω υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα και για μένα αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά ανησυχητικέ. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποιες παραπάνω πληροφορίες για την κατάσταση στην Κροατία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γεννάκου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερω ε, <clears throat> όσου ήρθαν σήμερα στην ακρόαση ε, και έθεσαν πραγματικά με πάρα πολύ ρεαλιστικό τρόπο την ε, υπάρχουσα κατάσταση. Ε, είναι γεγονός ότι οι σχεδιασμοί γύρω από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές <coughs> δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γύρω από μια πραγματικότητα και κυρίως πολλές φορές δεν μπαίνουν στην διαδικασία για το πώς μπορεί να αναστραφεί αυτή η κατάσταση, πώς μπορεί να αλλάξει. Και είναι φανερό ότι για να αλλάξει τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Είναι εξαιρετικά δύσκολα. Ο τομέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη του την έκταση, από την ισότητα των φύλων, το τράφικινγκ των γυναικών και τα άλλα ζητήματα που εμπλέκονται, αλλά κυρίως οι εμπειρίες του πολέμου, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που και αν ακόμα εμείς δεν επρόκειτο να συνενέσουμε στο να γίνουν αυτοί μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ίσως δεν είναι στην πραγματικότητα έτοιμες ορισμένες χώρες από αυτές να γίνουν μέλη, θα είχε σημασία για την Ευρώπη στα πλαίσια της, ε, του τομέα της ανάπτυξης για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά ε, στο να επιταχυνθούν ορισμένες διαδικασίες. Το ζήτημα δεν είναι αν εξυγχρονίζει τη δικαιοσύνη. Είναι βέβαιο ότι οι νόμους έχουν περάσει. Δεν εφαρμόζονται. Είναι προφανές ότι δεν εφαρμόζονται. Δεν υπάρχει στη συνείδηση του λαού η αντίληψη, γι' αυτό και γίνονται οι επιθέσεις του δημοσιογράφου. Και αυτό είναι ένα ερώτημα για τους προσκεκλημένους μας. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα και αποτελεσματικότερα. Γιατί είναι γεγονός, το είπε ο κύριος Ζέμπεκ, ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα, των οποίων το αποτέλεσμα εγώ έχω αμφιβολίες αν είναι ε, θετικό στο βαθμό που έπρεπε και νομίζω, κυρία Πρόεδρε, αυτό πρέπει να αναζητήσουμε και σε επόμενες συνεδριάσεις μας με το αντικείμενο αυτό θα βοηθούσαμε ουσιαστικά, νομίζω, ε, και τους ανθρώπους εκείνους και ε, εάν ε, θέταμε ως ισχυρότερο όρο τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρα από τα κριτήρια της Κοπενχάγης ως αρχικό και βασικό στοιχείο για την οποιαδήποτε διεύρυνση της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου. Κάνω την, επόμενη, ε, την ακόλουθη πρόταση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ματζίρσινγκ της Διεθνούς Αμνηστίας και μετά ε, ε, τις τελικές παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντού Μιρέλ και θα δώσω και το λόγο στον κύριο Κούπαν σαν επικεφαλής αντιπροσωπείας για να σχολιάσει όσα ακούσαμε. Δεν ε, ξεχνώ ότι έχουμε μία ομάδα βουδιστών ε, μοναχών ε, από το Βιετνάμ στο βάθος της εθούσης οπότε δύο λεφτά διαθέστε τους να μας πούν τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Ουσιαστικά ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια και το οποίο σχεδόν ξεχάσαμε σήμερα, γι' αυτό ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αναφέρουμε το, στο θέμα των γυναικών που βιάστηκαν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη κατά τον ε, ε, πόλεμο διότι έχω εδώ ένα αντίγραφο και όποιος θέλει μπορώ να του το δώσω παρά ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να ε, συζητήσουμε ε, διότι υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες ε, βιάστηκαν κατά τον πόλεμο χωρίς να έχουν πρόσβαση ή στη δικαιοσύνη κατά αυτών των βιασμών και επίσης δεν υπάρχει και κοινωνική αποκατάσταση για αυτά τα εγκλήματα. Όταν μιλώ για έλλειψη δικαιοσύνης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κατά τη διάρκεια του πολέμου όλοι συζητούσαν για τα προβλήματα αυτά και μιλάμε για ένα αριθμό μεταξύ 20 και 50 χιλιάδων γυναικών που βιάστηκαν κατά τον πόλεμο και η IC2I ε, μόνο παραπέμψει στη δικαιοσύνη 18 περιπτώσεις για σεξουαλική βία ε, και ορισμένα ε, ισότιμα 12 μάλλον έχουν προσαχθεί από τη Βοσνία Ερτσεγοβίνη Μιλάμε για 30 περιπτώσεις και παραμένουν πάρα πολλές οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί από κανέναν. Όπως γνωρίζετε, οι δράστες αυτών των εγκλημάτων ε, ε, κινούνται ελεύθερα στη Βοσνία Ετζεγοβίνη και ενδεχομένως αποφασίζουν και τη μοίρα των επιβιωσάντων ε, από ό,τι πληροφορούμαστε. Ε, οι γυναίκες αυτές ήταν φτωχές στην Υπεθρό χωρίς απασχόληση, χωρίς ψυχολογική στήρεξη, είναι τραυματισμένες, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτών των γυναικών. Μιλάμε επίσης για συμφιλίωση, διότι οι γυναίκες αυτές ε, δεν μπορούν να ε, επανέλθουν διότι οι βιαστές τους κινούνται ελεύθερα. Ε, όπως ξέρετε, όπως μας είπε και ο κύριος Χιμανίτσοβιτς, υπάρχει μεν το δικαστήριο όπου έχουν κριθεί περιορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν διεθνείς ε, δικαστές ε, και εισαγγελείς αλλά αυτή τη στιγμή μάλλον η εντολή των ε, διεθνών δικαστών λύγει τον επόμενο μήνα και δεν υπάρχει καμία στρατηγική για τις περιπτώσεις αυτές τις οποίες έχουμε παρακολουθήσει τόσο καιρό. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Μπορούμε να εξασκήσουμε πίεση ε, να ε, επεκταθεί η εντολή των δικαστών αυτών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και είναι κρίσιμο διότι χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να αναφέρω είναι ότι μπορείτε να επιμείνετε από τις αρχές της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, να συνδράμουν τις γυναίκες αυτές οι οποίες ε, ε, βιάστηκαν κατά τον πόλεμο να μπορέσουν να βρουν δουλειά, να έχουν ψυχολογική στήριξη. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν μέσω της υιοθετήσεως μιας στρατηγικής και επιλύσεως των προβλημάτων για να υπάρξει και κάποια αποζημίωση. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θα παρακαλέσω τον κύριο Μιρέλ τώρα να απαντήσει και ίσως ε, να απαντήσει τι έχει να πει για τις ε, επιβιώσαντες από ε, τους βιασμούς αυτούς. Ίσως δεν θα απαντήσω κατά σειράν, θα ξεκινήσω με την παρατήρηση της κυρίας Γιαννάκου ότι έχει δοθεί ε, σημαντική οικονομική στήριξη και ποια ήταν η έκβαση. Βεβαίως υπήρξε μεγάλη οικονομική στήριξη, πολύ σωστά νομίζω, για την ε, ε, στήριξη των εθνικών δικαστηρίων και διαφόρων παραμέτρων που αναφέραμε αλλά υπάρχουν τόσες ανάγκες όταν έχετε χιλιάδες περιπτώσεις οι οποίες ακόμη εκκρεμούν στα δικαστήρια οι οικονομικοί πόροι που χρειάζονται είναι περισσότεροι και θα χρειαζόμαστε και περισσότερους εισαγγελείς, περισσότερους δικαστές. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει διατεθεί σωστά η χρηματοδότηση, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους πόρους. Και ακόμη πιο σημαντικό από την ε, χρηματική βοήθεια είναι η πολιτική θέληση στις χώρες αυτές να επιταχύνουν τη διαδικασία, να ε, διαθέσουν ε, περισσότερους πόρους στην δικαιοσύνη, να συμφωνήσουν εις, ε, τις εκδόσεις από τις χώρες αυτές και δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα οικονομικό. Η ερώτηση του κυρίου Πρόντι. Νομίζω ότι εάν υπήρξε ένας πόλεμος στα Βαλκάνια δεν μπορούμε δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα αποκατασταθεί η πρώην Ιουγκοσλαβία εκτός και αν παρανόησε αυτό το οποίο είπατε. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι σε κάθε χώρα να αναλυφθούν πολύ πιο σοβαρές προσπάθειες δικαστικής μεταρρύθμισης ε, αντιμετωπίσεως ε, της ε, επιστροφής των προσφύγων, επιλύσεως της κατάστασης των βιασμών και να υπάρξει μία πραγματική περιφερειακή συνεργασία η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά συνέδρια, θαυμάσιες δηλώσεις, αλλά η μόνη συνεργασία την οποία διαβλέπουμε είναι όταν συμφωνήσουν διάφορες κυβερνήσεις να βοηθήσουν τη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΠΑ για να ξεκινήσουν ορισμένα προγράμματα. Χρειάζονται όμως και πολλά ακόμη. Τρίτον, η ερώτηση του κυρίου Ζέμ και για την Κροατία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι υπήρξε ε, πρόοδος στην ε, Κροατία και η, ε, χάρη στην ε, διαδικασία προσχωρήσεως έχουν ξεκινήσει πολλά προγράμματα αλλά όπως σας είπα ε, η περιφερειακή διάσκεψη που ζήτησε η Σερβία επιβάλλεται για να μπορέσει να έχει μία αίσια έκβαση και πιστεύω ότι όλοι οι δωρητές θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν οικονομικά κατά κάποιον τρόπο. Όσον αφορά την ερώτηση ή μάλλον τον αριθμό των ερωτήσεων που έθεσε η κυρία Ντεκάιζερ. Καταρχήν, όσον αφορά την αποστολή στο Κωσυφοπαίδιο, αν θυμάμαι καλά Φεβρουάριο-Μάρτιο ε, φέτος ε, η ε, αποστολή έχει πλήρως ε, εγκατασταθεί και μπορεί να παρέμβει. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μία σειρά περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου όπου έχει βγει απόφαση του δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου, άρα έχει γίνει σωστή δουλειά, αλλά σε θέματα δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι αν σήμερα καθαρίσουμε έναν δικαστή ή έναν εισηγητή ε, μπορούμε να έχουμε και τις αποφάσεις. Έχουμε περίπλοκους φακέλους, χρειάζεται περισσότερος χώρος, χρόνος από ό,τι σε άλλους τομείς, αλλά πιστεύουμε ότι η αποστολή αυτή θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο και όπως είπε και η κυρία Τζόνς ξεκινήσαμε με τους εξαφανισμένους ανακοινήσαμε το θέμα αυτό ε, ψάξαμε στα, ε, στις διάφορες ιστοσελίδες έχουμε ξανανοίξει τους φακέλους, χρηματοδοτούμε ε, αν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδοτήσεως για την αναζήτηση ε, των πτωμάτων και υπάρχει μία αντίληψη αρνητική της κοινή γνώμης για τα Βαλκάνια. Οι χώρες δεν συμφωνούν, υπάρχουν ακόμη διμερείς ε, συμφωνίες και διαμάχες και όπως είπαμε και στο έγγραφο στρατηγικής. Γι' αυτό το λόγο τα θέματα αυτά των μειονοτήτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ βασικό για κάθε ε, χώρα των Βαλκανίων να εργαζόμαστε σοβαρά για να επιλύσουμε τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Μιρέλ. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί τώρα η ακρόασή μας και θέλω να δώσω το λόγο εις τον κύριο Κούκαν, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ σύντομα γιατί είμαστε πιεσμένοι από το χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλοξενούμενους που ήρθαν και εμπλούτησαν με τις γνώσεις τους και τις πληροφορίες τους στη συζήτηση. Πιστεύω ότι η παρουσίαση του κυρίου Σέμπεκ ήταν πολύ θετική και με αυτή την ευγλωτία μπορούμε να προχωρήσουμε αλλά θα ήθελα να πω ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια πραγματική περιοχή με πραγματικό κόσμο που ζουν μια πραγματική ζωή, που αναπτύσσονται και αξίζουν τη βοήθειά μας, την στήριξή μας και τη συνεργασία μας όσο και να είναι διαιρημένη θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μην περιμένουμε 800 χρόνια για να τους προσφέρουμε δημοκρατία και να τους δεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τον κύριο Μιρέλ, νομίζω ήταν πολύ επίκαιρες οι παρεμβάσεις σας και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευχαρίστως θα συνεργαστεί όπως είπατε ούτως ή άλλως υπάρχει στήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα ε, εκπεραιώνει ένα ψήφισμα ε, για ε, την στρατηγική διεύρυνση βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής που συζητήθηκε στις εξωτερικές υποθέσεις και νομίζω το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο θα υιοθετηθεί το ψήφισμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Είστε, η πρόεδρος είναι πολύ αυστηρή η συζήτηση απέδειξε το τη σοβαρότητα αυτής της Επιτροπής. Η κυρία Γιαννάκου, η κυρία και Ντεκάιζερ έκαναν πολύ σοβαρές και πολύ επίκαιρες ερωτήσεις και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για, αυτή την, ε, εξαιρετική, για τις εξαιρετικές τελικές παρατηρήσεις. Θα ξανασυζητήσουμε το θέμα ε, προσεχώς και σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες σας προτάσεις από τον οποίο θα δουλέψουμε. Και τώρα είναι δικαίωμα και καθήκον μου να πω στους διερμηνείς ότι η επίσημη συνεδρίαση ολοκληρώνεται, εμείς θα συνεχίσουμε μερικά λεπτά στα αγγλικά. Χαίρετε. Λοιπόν. It's a delegation from uh, Plume Village Monastery from France, if I understand well